Good morning Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλους τους α, επισκέπτες μας. Καλώς ορίζω και τους ευρωβουλευτές, σημερινή συνεδρίαση. Βλέπω ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ομάδα όμορφων ανδρών και γυναικών, που είναι αστυνομική από την Ιταλία. Και ο πατέρας μου ήταν αστυνομικό και αισθάνομαι μέσα στο σπίτι μου. Χαίρομαι που σας βλέπω μπροστά μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι. Να συνεχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας από χθε. Έχω κάποιες ανακοινώσει να σα κάνω καταρχήν. Ορισμένες δεν θα σα ενδιαφέρουν όλους, αλλά πρέπει να γίνουν με βάση του κανονισμού μα. Χθε οι συντονιστέ ε, πήραν τι εξή αποφάσεις ε, υιοθέτησαν την ε, ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου και όλες, όλα τα αιτήματα της ομάδας ε, για την ατζέντα του Φεβρουαρίου ε, λήθησαν υπόψη. Η αναφορά 224 του 2018 που αφορά τους ε, δημοσίους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων θα συζητηθούν ε, στο εργαστήρι για την, το θέμα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων στις 2 Απριλίου. Και θα προσκαλέσουμε και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Διάφορες ε, αναφορές θα διαγραφούν από την ατζέντα του Φεβρουαρίου, όπως ζήτησαν οι ομάδες, για το 20, σημείο 29. Η ομάδα, οι ομάδες ζήτησαν από τη Γραμματεία να δουν τι θα γίνει αν μπορούν να προσθεθεί στη μερίσια διάταξη και το θέμα κάποιο, για κάποια οικονομικά ζητήματα. Επίσης, ένα σύντομο ψήφισμα ε, για την ε, διαχείριση αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λάβουμε υπόψη όλες τις σχετικές αναφορές με το θέμα αυτό και θα τις ε, στείλουμε στην ε, διάσκεψη των Προέδρων προς έγκριση ή απόρριψη. Ε, το ΕΛΚ ζήτησε να αναβληθεί το σύντομο ψήφισμα, ε, που ζήτησε να αναβληθεί το, ψήφι, να αναβληθεί, συγγνώμη, το σύντομο ψήφισμα, απορρίφθηκε. Επίσης, έχουμε τέσσερις ακόμα συνεδριάσεις πριν λήξει αυτή η θητεία και θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα για τις αναφορές στη γραμματεία για τις αμφισβητούμενες συστάσεις. Οι περισσότερες συστάσεις μου ακολουθήθηκαν εκτός από την 0758 και 0760 που θα παραμείνουν ανοιχτέ. Και τα σημεία 335 ε, και το 318 θα παραμείνουν ανοιχτά. Επίσης, ε, καταγράψαμε το σχέδιο προγραμματός της ακρόασης για την κλιματική αλλαγή και την άρνηση της κλιματικής αλλαγής και συμφωνήσαμε ότι η Γραμματεία θα επιλέξει τους ε, υποψήφιους ομιλητές ανάλογα με το κατά πόσο είναι διαθέσιμοι για να έρθουν στο, στην εκδήλωση. Ε, πρόταση του, των σοσιαλιστών για το ελεγκτικό συνέδριο ε, για να, παρακολουθ... να δώσουμε συνέχεια στην προηγούμενη μελέτη που είχε εκδώσει το ελεγκτικό συνέδριο για το... την ενωσιακή νομοθεσία και ε, απορρίφθηκε η αίτηση για να ξανανοίξει, να η αναφορά 636. Αυτά αποφασίσαμε χθες. Τώρα πάμε στην ψηφοφορία. Θέλω συνάδελφοι να ακολουθήσω το παράδειγμά μου. Βγάλτε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας, βάλτε τις στο μηχάνημα. Θα ψηφίσουμε για το αποτέλεσμα της ε, Επιτροπής Αναφορών, ε, τα των συζητήσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Απορρίπτεται. Κοιτάξτε μας πώς απορρίφθηκε. Πολύ ε, βραχία κεφαλή απορρίφθηκε. Το δεύτερο τμήμα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 κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 έχει αποσυρθεί 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίσμα τώρα Πέρα οφορία με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ψηφοφορία, ε, πλειοψηφία απορρίφθηκε. 15 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 17 με μια προφορική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Απορρίπτεται. 19. Όχι, ελέγχουμε πρώτα ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Εδώ. Δεν ψηφίσατε όλοι ακόμα. Ωραία, τώρα πέρα. Τη απορρίφθηκε. Όντω. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές την ελέγχουμε επίσης ηλεκτρονικά αυτήν δεν έχουμε δεν είμαστε πολλοί πάλι απορρίπτεται πάλι με τον ίδιο τρόπο την ίδια πλειοψηφία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 έχει αποσυρθεί. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά να ελέγχουμε καλύτερα. Απορρίπτεται, ούτω ή άλλω. Πίτερ, καλή τύχη την επόμενη φορά. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Θέλετε να ελέγξετε την, την 34. Λοιπόν, την ελέγχουμε χρονικά 34. Απορρίπτεται. Άρα, μια και ψηφίσαμε 36, πάμε στη 35. 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική ψηφοφορία για την 37, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα καταπίπτει. Και πάμε στο 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. 42. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος και στο επόμενο. 8-8 απορρίπτωται. Το 44 απορρίφθηκε. Επομένως, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 43. Επίσης χωριστή ψηφορία το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Ζητείται ηλεκτρονικός έλεγχος. Μάλιστα λέει Το πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα επίσης. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πρέπει όλοι να ψηφίσετε. Ακόμη ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως προσωπικά μια που ήμουν η συγγήτρια. Ε, και τώρα προχωρούμε. Συνάδελφοι, αν θέλετε να φύγετε, παρακαλώ να το πράξετε ταχαίως και ησύχως, λέει ο Πρόεδρος.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 Now when people have left the room. Μια που απεχώρησαν αυτοί που ήθελαν, πάμε τώρα στην Ερευνητή των Πραγμάτων Ευρωπαϊκής, στο Βαλεντρό της Ιταλίας. Αυτό έγινε τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές. επικεφαλής ήταν ε, η Μπιατρίς Μπεθέρα, στην οποία θα της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε μισό λεπτάκι να περιμένω για να καθίσουν οι συνάδελφοι. Είναι τιμή μου να σας κάνω αυτόν τον απολογισμό της αποστολής. Πρόεδρος, νομίζω το είπα, το είπα ευγενώς πριν από μισό λεπτό. Όποιος δεν προτίθεται να μείνει, να αποχωρήσει ήσυχα και με τρόπο κομψό, ούτως ώστε να μην γινόμαστε ρεζίλ μπροστά σε όλους αυτούς τους αστυνομικούς τους προσκεκλημένους εννοεί η Πρόεδρος προφανώς. Α, τώρα βλέπω ότι συχάσατε, συγκεντρωθήκατε. Οπότε, Μπιατρίς, για άλλη μια φορά προσπάθησε να μας τα πεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ε, ε, επισκέπτες μας που μας δίνουν τόση ασφάλεια και ακριβώς αυτή η, η, αποστολή αφορά τη χώρα του στην Ιταλία και ε, για μένα από όλες τις αποστολές που έκανε σε αυτή τη θητεία. Αυτή ήταν μία από τις ε, πιο θετικές, πιο παραγωγικές, από τις καλύτερα οργανωμένες. Ε, πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά όσον αφορά την επιτυχία αποτελεσμάτων και όσον αφορά την ε, πρόταση του Κοινοβουλίου για κάτι συγκεκριμένο. Να υποστήξετε το Κοινοβούλιο για συγκεκριμένο πρόβλημα συγκεκριμένους ανθρώπους. Επίσης ευχαριστώ τους συναδέλφους που με συνόδευσαν γιατί ε, τα έκαναν όλα πάρα πολύ εύκολα η Ελεονόρα. Ε, διάφοροι τέλος πάντων, δεν ξέρουν όλοι εδώ, ούτε η Άννα Μιράντα, τέλος πάντων. Και όπως λέγαμε, στις 17 και 18 λίγο πριν τα Χριστούγεννα κάναμε αυτή την ε, αποστολή, αυτή την επίσκεψη για να ερευνήσουμε κάποια πράγματα στο Βαλεντόρα του Πεδεμοντίου στην Ιταλία και πήγαμε στο Λιτσακάστελ στην Καμπάγια, κάποιους δήμους δηλαδή και το πιο βασικό σε αυτή την αναφορά και σε όσες προηγήθηκαν για το θέμα ήταν το εξής. Να δούμε πώς κάποιος έκανε αυτή την αναφορά. Πρόκειται για έναν δήμαρχο. Αυτό δείχνει το πόσο ενδιαφέρονται οι Ευρωπαίοι και αυτός ο δήμαρχος κατάφερε να συσπυρώσει πάρα πολλούς πολίτες, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, από διάφορα θεσμικά όργανα, από το δικό του Δήμο και από άλλους. Και όλοι αυτοί με αποφασιστικότητα, με επιχειρήματα ισχυρά, ε, έκαναν κάποια κατάθεση ε, όσον αφορά το θέμα τους και ήρθαν εδώ επανειλημμένα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκαν και την ε, Δευτέρα το απόγευμα είχαμε μία ακρόση τέσσερις ώρες και βάλε και ήρθαν διάφοροι ομιλητές και μας είπαν τι γίνεται με όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την αναφορά και ήρθαν όπως είπαμε από πανεπιστήμια, από θεσμικά όργανα, ήρθαν πολίτες από κάποιους φορείς ε, πολιτιστικούς, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της, της ε, περιφερειακής διοίκησης και φυσικά από τον ίδιο τον ε, Δήμο. Βέβαια, δυστυχώς δεν υπήρχε και έλλειψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεν απάντησε στην επιστολή μας. Δεν ε, μας έστειλε καν την τοποθέτησή του. Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε ζητήσει, αλλά και ο ίδιος ο αναφέρον. Την επόμενη μέρα πήγαμε επί τόπου. Πήγαμε να δούμε τι γίνεται εκεί, στις εγκαταστάσεις που αφορούσε η αναφορά. Μας, μας είπαν εξαντλητικά ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε τα είδαμε και όλα επί τόπου. Επομένως, ε, μετά από την εξαντλητική παρουσίαση, ήταν εξαντλητική και η δική μας ε, έκθεση των πεπραγμένων και είδαμε ότι θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί Υπάρχει πρόβλημα εκεί όσον αφορά τις αποχετεύσεις, υπάρχει τις, τις χωματερές και για τα επιφανειακά ύδατα και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα μέτρα. Επίσης, άλλο συμπέρασμα, προφανές, ο συντονισμός μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Το κράτος, η περιφέρεια, τοπικέ αρχές είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για τον Ελλάδα. Μόνο ε, ένα κομμάτι της διοίκησης, ένα επίπεδο της διοίκησης. Ε, βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από κάποιο κράτο μέλο να εφαρμόσει, να μεταφέρει στο ιστορικό δίκαιο την οδηγία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει το κράτο. Δεν υπάρχει έναρξη διαδικασία παραβάσεω. αλλά είπαμε ότι δεσμεύτηκαν σε αρχές να πάρουν κάποια διαδροτικά μέτρα και να μην έχουν τα ίδια προβλήματα στο μέλλον. Ε, Επίση ούτε να υπάρξουν στην ε, Βαλεντόρα ή αλλού στην Ιταλία τέτοιου είδου χωματερέ γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ ε, ε, έντονο το πρόβλημα στο τώρα ε, Είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, αλλά δεν είναι μια περίπτωση μοναδική, ούτε καν για όλη την Ιταλία. Είναι συστημικό το πρόβλημα στη χώρα και αλλού. Επομένως, εμείς θα πρέπει κάτι να κάνουμε, να έχουμε κάποια θέση κρυστάλλινη Οπότε επί τη βάση του σχεδίου κειμένου που έχουμε ε, θα τα πούμε ξανά τον Μάρτιο, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι συστάσεις για λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι να ισχύσει αρχή της πρόληψης, επιμέλειας κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το timing. Το τι θα γίνει από 1η Φεβρουαρίου Γι' αυτό, όπως είπε και χθες η κυρία Εύη, θα πρέπει να δούμε αν γίνεται ψήφισμα στην Ολομέλεια σχετικά. Κύριος και μέλο, ο Δήμαρχος του Τανσάνο, συνάντησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος στις 15 Ιανουαρίου, μετά την ε, αποστολή μας. Και από ό,τι γνωρίζουμε μετά από αυτή την ε, συνάντηση συνέχισε την αυστηρή του θέση όσον αφορά την πολιτική του Υπουργείου. Πάντως η επίσημη θέση του Υπουργείου παραμένει κατά κάποιο τρόπο ε, μια θέση που δεν καλύπτει τι ευθύνε που θα έπρεπε να έχουν αναλάβει. Θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να επιληθεί το πρόβλημα. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των σχετικών οδηγιών, των σχετικών με αυτή την αναφορά. Τα υπόλοιπα μπορούν να σας τα πούνε βέβαια και οι συνάδελφοι που ήρθαν στην αποστολή. Πάντως και πάλι ευχαριστώ για την ευκαιρία να πάω για αυτή την ερευνητική αποστολή αλλά ήταν επίσης ε, πάρα πολύ επαγγελματική υποστήριξη το έργο των συνεργατών μας της Επιτροπής Αναφόρων ήταν η βοήθειά τους ε, πάρα πολύ πολύτιμη η Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε Πρόεδρος Επιτροπής που ανέλαβε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που ηγηθήκατε της ε, αντιπροσωπείας για την επίσκεψη. Μικρή αντιπροσωπεία, αλλά η οποία απηχούσε την ε, πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου από όλα τα κόμματα. Ε, ο κύριος Κύριο, ε, ε, άλλοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, βεβαίως η κυρία Έλλη, Εύη μάλλον, συγγνώμη, εσείς βεβαίως η ίδια. Άρα ήταν μια θαυμάσια σύνθεση, ισορροπημένη και αναμένω με ενδιαφέρον την συζήτηση, την συνεδρίαση μάλλον του Μαρτίου, όπου θα συζητήσουμε την έκθεση, την οποία ήδη περιγράψατε. Θα ήθελα τώρα να ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συμφωνείτε. Α, πρώτο, πρώτο κύριος Πέτερ Γιάρ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μικρό σχόλιο. Ήταν ε, πραγματικά θαυμάσια η προετοιμασία. Ανταποκρινόταν ακριβώς ε, και στις δικές μας ιδέες καλά και σφιχτά οργανωμένη. Ευχαριστώ βεβαίως και τη Γραμματεία αλλά και τους συναδέλφους ε, που έδρασαν επί τόπου. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα ταξίδι στο παρελθόν. Η διαχείριση αποβλήτων μου θυμίζει ιστορίες που έχουμε ζήσει από το 1970 και μετά και μου φαίνεται καλό ότι οι δήμαρχοι λένε stop, ως εδώ και μη παρέκει. Οι ορισμένοι προτείνουν απλές λύσεις, θα, πάρουμε εγκαταλειμμένα λατομεία και θα τα γεμίσουμε με τα απορρίμματα. Εκεί χρειάζεται κάποια αντίδραση και κάποια αντίσταση. Θα μας απασχολήσει επαρκετόν η συγκεκριμένη αναφορά. Ήδη η απουσία εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης από την ε, αποστολή, από την επίσκεψη δηλαδή, την εξεταστική επίσκεψη, δείχνει ότι δεν είναι στην ημερήσια διάταξη της κεντρικής διοίκησης το θέμα. Χρειάζεται να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, την ε, τοπική κοινότητα, χρησιμοποιούν τεχνολογία του περασμένου αιώνα. Υπάρχουν καλύτερε τεχνολογικές λύσεις είναι λίγο δύσκολο. Ε, δηλαδή, οι πολίτε μπορούν να, να μπορούν να πούν όχι. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να προτείνουν οι ίδιοι λύσει ή πάντω όχι αναγκαία. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια στρατηγική δράση από την κεντρική κυβέρνηση, διότι χρειάζεται μια συνολικότερη αντίληψη δράση. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει από το κέντρο, διότι οι τοπικέ κοινότητε βρίσκονται ω τελευταίο κρίκο τη αλυσίδα. Άλλωστε στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα χρειαστεί να εγκύψουμε στο θέμα αυτό με ιδιαίτερη έμφαση και παρακαλώ και τους και τις υφιστάμενες συναδέλφους, ιδίως Ιταλών, μην αφήσετε τη Ρώμη να ξεφύγει, την πρωτεύουσα δηλαδή, να ξεφύγει από τις ευθύνες τις οποίες οφείλει να αναλάβει χρειάζεται μεγάλη και διαρκή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ήδη, ήδη έχουμε κάπως καθυστερήσει. σα παρακαλώ να είστε συντομότατοι. Η Ελεονόρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω οπωσδήποτε να παρέμβω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ την κυρία Πεσερέλ για την έκθεσή της. Ευχαριστώ τους αναφέροντες ε, που έθεσαν αυτό το θέμα εγκύπτει από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αναφορά, γιατί ακούτε πραγματικά τα προβλήματα που προέρχονται από τι κοινότητε μα, του Δήμου μα. Εγώ ως Ιταλίδα προέρχομαι από, την, ε, από κοντινή εκλογική περιφέρεια και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι είναι ένα θέμα για το οποίο η εθνική κυβέρνηση της Ιταλίας πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ας μην ε, κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Α μην κρύβουμε το κεφάλι στην άμμο. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτούς τους ε, δημάρχους που επί χρόνια μάχονται. Το θέμα της ε, διαχείρισης των αποβλήτων είναι δύσκολο και ευαίσθητο θέμα να αντιμετωπίσουμε και στην Ιταλία αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Και χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική μετάβαση προς την ε, κυκλική οικονομία και στην αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η λύση που προτείνεται το να ανοίξουμε νέες χωματερές δεν είναι η ευκταία λύση. Όταν μπούμε στην ουσία της έκθεσης ε, θα πούμε ιδέες, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε φυσικά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και το θέμα της, ε, του γεωλογικού φραγμού των χωματερών πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά πρέπει να ε, σεβαστούμε και, και να εφαρμόσουμε σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ λοιπόν τη συνάδελφο για την, ε, τα όσα μας είπε. Περιμένω να δω το έγγραφο, να δω πώς θα συνταχθεί για να μπορέσουμε να εργαστούμε επικοδομητικά επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε και εγώ ξεκίνησα την συνάντηση λέγοντας ότι αποφάσισαμε χθε να συντάξουμε σύντομο ε, ψήφισμα για την διαχείριση των αποβλήτων και αυτό θα αποτελέσει και τον πυρήνα το ψηφίσματο μαζί με άλλα παρόμοια θέματα που σημειώνονται σε άλλε χώρε μέλη. Μάλιστα, τώρα α αναμείνουμε να δούμε το έργο που θα κάνουμε με βάση την ίδια την έκθεση. Ευχαριστώ όλες και όλους για την καρποφόρο αυτή και επιτυχημένη επίσκεψη και ας περάσουμε στο επόμενο που είναι το υπαριθμό 14. Το υπαριθμό 14 που όπου πρόκειται για τρεις διαφορετικές αναφορές και οι τρεις αναφέρονται στις ε, τοπικές αστυνομίες που δεν εντάσσονται στις ε, ε, βασικές αστυνομικές δυνάμεις της, του Ιταλικού κράτους. Έχουν και διαφορετικό καθεστώς από την Εθνική Αστυνομία. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό θέμα. ευχαριστώ να δώσω τον λόγο στον κύριο Λουίτζι Μαρούκι και στον κύριο Φραντσέσκο Γκαρόφαλο και θα τους δώσω το λόγο για πέντε λεπτά και ακολούθως ο επόμενος αναφερόμενος που έχω τα αρχικά του, PB και τέλος του Μάριο Ασιρέλη. Θα παρακαλέσω να είστε σύντομοι για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων Ευρωβουλευτών. Πρώτα η κύριοι Μαρούκη και Γκαρόφαλο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ είναι η πρώτη φορά που μιλάω εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν μια πρώτη φορά που μας φέρατε εδώ και δεύτερον ε, γιατί μου δώσατε το λόγο. Ε, εκπροσωπούμε την Ιταλία, ε, ερχόμαστε από το Παλέρμο και το Τωρίνο. Ε, εκπροσωπούμε 60.000 ε, δημοτικούς αστυνομικούς της Ιταλίας που είναι πραγματικοί αστυνομικοί, αλλά έχουν μια σύμβαση που τους εξισώνει με τους υπαλλήλους των Δήμων. Έχουμε ίδιο μισθό με τους υπαλλήλους αυτούς και έχουμε μηδενική προστασία. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή σας τουλάχιστον να παρέμβει, να πιέσει την Ιταλική κυβέρνηση, ούτως ώστε να δώσει αυτούς τους 60.000 άντρες Φυσική προστασία, παραδείγματο χάρη αλεξίσφαιρο γυλαίκο και κράνος κατάλληλο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Δύο δημοτικοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν λόγω έλλειψης προστασίας. Έχουμε διατάγματα τα οποία εξέδωσαν δύο, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία. Ε, πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, είμαστε παρόντες σε όλη την Ιταλική επικράτεια. Ε, η δραστηριότητά μας είναι 100% αστυνομική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουμε εργαλεία προστασίας. Το 2018 200 ε, δημοτικοί αστυνομικοί ε, έτυχαν, έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης. Ε, και αντιμετώπισαν και πολλοί άλλοι προβλήματα υγείας. Αυτά τα πράγματα δεν τα λέμε για πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήρθαμε το 2017 και μιλήσαμε για αυτά. Ζητήσαμε από την Επιτροπή σας να παρέμβει και να μιλήσει στην Ιταλική κυβέρνηση. Ε, στο Υπουργείο Εσωτερικών στείλατε μία επιστολή, Πρόεδρε, και το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο από το επιθυμητό. Γιατί το Υπουργείο ε, αποφάσισε ότι είμαστε υπάλληλοι των Δήμων και Κοινοτήτων και απλώς αστυνομεύουμε παράλληλα ως τέτοιοι υπάλληλοι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στον κόσμο. Ή είμαστε αστυνομικοί, ή είμαστε δημοτικοί υπάλληλοι. Ή θα είμαστε αστυνομικοί με την προστασία που έχουν όλοι οι αστυνομικοί όλου του κόσμου ή αλλιώ θα είμαστε υπάλληλοι α πούμε των Δήμων και Κοινοτήτων. Πάμε το πρωί χαλαρά και γυρνάμε το βράδυ σπίτι χαλαρά. Άρα δεν δουλεύουμε το βράδυ κτλ. Δεν παρεμβαίνουμε εκτό ωρών εργασία. Εμεί είμαστε όμως παρόντε 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 60 θύματα. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί, η εθνική αστυνομικοί, ας πούμε, το, της Ιταλίας, ε, δεν είχαν ούτε ένα θύμα. Γιατί εμείς είχαμε 60 ε, θύματα οι οποίοι α, ποδοπατήθηκαν από αυτοκίνητα, ε, τους α, πυροβόλησαν κτλ. Ή πέσανε θύματα εγκληματιών. Ε, Νομίζω ότι η Επιτροπή σας να ακούσει αυτά που είπαμε και στην πρώτη ακρόαση και να επιμείνει μετά την άσχημη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών να, κάνετε, να έρθετε στην Ιταλία, να κάνετε μια επίσκεψη, να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τι κάνουν αυτοί οι άντρες, οι οποίοι εκπροσωπούν τον νόμο. Αναφέρονται στο Ιταλικό Σύνταγμα. Στην πραγματικότητα τους χρησιμοποιούν οι θεσμοί για τη μαύρη τους δουλειά. Τους βάζουν να κάνουν μαύρη εργασία τα επίσημα θεσμικά όργανα. Δεν έχουμε καμία προστασία, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας ακούσατε. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που ανήκουν σε αυτή την Επιτροπή. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ζητάω ταπεινά να δείτε τι, τι πραγματικά συμβαίνει. Να στείλετε μία αντιπροσωπεία από ευρωβουλευτές στην Ιταλία. Για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τι συμβαίνει και τι δουλειά κάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρησιμοποίησατε τα πέντε λεπτά σας. Υπάρχει τώρα άλλος αναφερόμενος, τα αρχικά του οποίου είναι πι Και τον παρακαλώ. Α, είναι ο Γκαρόφαλο. Okay, one minute. One minute. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι τώρα να συμπλώσω κάτι σε αυτό που είπε ο ο Πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε κάποια πρόοδο στη χώρα μα, αλλά και γενικότερα σε όλε τις χώρε τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ότι για όλες τις προσπάθειες γίνονται σε όλες τις πόλεις Ιταλίας είναι η τοπική αστυνομία. Όμως έχουμε δεχθεί τώρα πλήγματα. Και έχουμε πάρα πολλέ αρμοδιότητες, αλλά είμαστε τώρα στο επίκεντρο αυτού του προβλήματος. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε, γιατί το έγκλημα έχει αυξηθεί. Και ε, έχουμε μόνο στα ίδια καθήκοντα με την εθνική αστυνομία, εμείς ως τοπική αστυνομία. Γι' αυτό και θέλουμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας και όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα πρέπει να δούμε οποίος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Μιλούμε για 60.000 άντρες και γυναίκες που εργαζόμαστε χωρίς να έχουμε καμία κάλυψη, καμία εγγύηση να απολάβουμε κάποιων στεγματικών δικαιωμάτων όποιος, όπως οποιοδήποτε υπάλληλο που εργάζεται στις άλλες αστυνομίες της ε, χώρας. Γιατί, ας πούμε, Ανά πάσα ημέρα μπορεί να είμαστε ε, εκτεθειμένοι σε κινδύνους και μπορεί να, να πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνουμε ενώ του καθήκοντος. Νομίζω ότι κατανοούμε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα, πλήρως το θέμα. Είχατε έρθει και παλαιότερα, σχετικά πρόσφατα. Το συζητήσαμε και τότε, επανέρχεσαι τώρα, να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα. Αντιλαμβανόμαστε το θέμα, το γνωρίζουμε και το mm. κατανοούμε καλά. Α έρθουμε τώρα στην δεύτερη ε, αναφορά που είναι υπαριθμών 93. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια παρουσίαση PowerPoint. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε και εσείς κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Βλέπετε ε, ότι στην πρώτη διαφάνεια λέμε ότι πρόκειται για λειτουργήμα και όχι απλώς μια εργασία. Φαίνεται όμως να μην λειτουργεί το... Α, το αρχίζει, ωραία από την ε, ρωμαϊκή ιστορία και μετά... Α, Ίσως πρέπει το ε, μηχάνημα αλλαγής των διαφανειών να έρθει λίγο πιο κοντά. Α, ίσως και απλώς δεν το γυρίσει τα ανάποδα, ναι. Να μιλήσουμε τώρα για τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει στείλει στην Επιτροπή Αναφορών και η επιστολή αυτή λέει για διοικητική αστυνομία που ασκεί ε, και ε, έρευνες για εγκλήματα, δεν μιλεί όμως για την προστασία των εργαζόμενων της Δημοτικής Αστυνομίας. Το πρόβλημα όμως είναι όταν οι πολίτες χρειάζονται ε, βοήθεια για κάποια, την αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού, είμαστε οι πρώτοι που ανταποκρινόμαστε. Έχουμε λοιπόν τα ίδια καθήκοντα και, τις, ε, και τους ίδιους κινδύνους. Τι γίνεται όμω με τι συλλογικέ συμβάσει εργασία. Όταν κάποιο εργάζεται ας πούμε σε μια τοπική ή ε, ε, κοινοτική αστυνομία, εκεί ισχύει το ιδιωτικό δίκαιο. Ενώ κάνει τα ίδια πράγματα όπω ε, όσοι κάθονται ας πούμε σε ένα γραφείο με πολύ χαμηλό κίνδυνο η διαφορά. Βλέπετε τι κάνουν ας πούμε οι λογιστές ε, των Δήμων και βλέπετε από την άλλη μεριά τι κάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί. 338 συλλήψεις το 2018. Άλλες αστυνομικές δυνάμεις και ε, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές έχουν διαφορετικές ε, συμβάσεις εργασίας. Και εκεί ισχύει το δημόσιο δίκαιο. Το ίδιο ισχύει, έχουν δηλαδή τους ίδιους κινδύνους αλλά με διαφορετική μεταχείριση. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία δική μου μετά από τέσσερις ώρες χειρουργείο που ε, είχα υποστεί ατύχημα. Είναι ε, εφιάλτης η υπόθεση αυτή για τις ε, τοπικές αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπαχθούμε στο δημόσιο δίκαιο. Και το πιο σημαντικό, εάν κάνει κάποιο λάθος η αστυνομία, οι τοπικές οι τοπικοί αστυνομικοί, αν τους βάλουν στη φυλακή δηλαδή, θα πάνε μαζί με τους απλούς ε, ε, κρατούμενους του ποινικού δικαίου. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για αυτούς. Άλλοι πηγαίνουν σε ε, φυλακή ειδική για αστυνομικούς και αυτό είναι το σωστό. Επίσης, πολλοί έχουν ήδη σκοτωθεί στην εκτέλεση του καθήκοντος. Θυμίζω την Σάρα Γκάμπαρο, η οποία ε, σκοτώθηκε στη διάρκεια ε, τροχαίου ελέγχου. Και άλλοι συνάδελφοι μου το ίδιο. Ο Νικολό Σαβαρίνο, ο οποίο ε, εφωνεύθη από εγκληματία στην άσκηση του καθήκοντό του. Ο Μικέλ Λιγκουρόρη, επειδή ε, πέθανε ο, διότι ε, εισέπνευσε τοξικά αέρια σε μια δραστηριότητα κατά της οικολογική μαφίας. Και ο Μάουρο Ντόντι, ο οποίος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε σημείο ελέγχου. Και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν απλώς τραυματιστεί την ε, αναφορά μας την υποστηρίζει η ε, περιφέρεια της Λομβαρδίας και ο έπαρχος. Έχει φτάσει η ώρα να ενηλικιωθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σας ευχαριστούμε πολύ και να είστε καλά. Πραγματικά θαυμάσια ε, παρουσίαση λέει η Πρόεδρος διότι ρίχνει φως στο γεγονός ότι πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη κατάσταση αυτή δηλαδή που συμβαίνει επί του παρόντος στην Ιταλία. Ας έλθουμε τώρα στον ε, Κλάουδιο Μάσκελα. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μάουρο Ασιρέλη. Ο Κλάουδιο Μασέλα είναι δίπλα μου. Ε, εκπροσωπώ και το συνδικάτο μας. Θα πρέπει να, δείτε ότι με βάση τον καονισμό ε, υπαχόμαστε σε διαφορετικό νόμο από τους υπόλοιπους αστυνομικούς. Οι τοπικοί αστυνομικοί ε, κάνουν και διοικητικά καθήκοντα, όπως και οι υπόλοιποι αστυνομικοί, αλλά και όλες τις άλλες δραστηριότητες της ε, ε, τροχέας, ε, της ε, δικαστικής αστυνομίας κτλ. Ε, προστατεύουμε το Δήμο και τις κοινότητες εναντίον των κινδύνων της δημόσιας ε, τάξης. Ε, επίσης προστατεύουμε και εναντίον των κινδύνων ε, που ε, είναι κατά της κοινωνικής ζωής. Ε, ζητάμε λοιπόν ε, να έχουμε την κατάλληλη προστασία. Ό, όσοι ανήκουν στην τοπική αστυνομία, όπως και η υπόλοιποι αστυνομικοί, παράδειγμα τους χάρη την Καραμπινιέρη, η εθνική αστυνομική η Guardia και Finanza κτλ. Ε, εξασφαλίζουν ε, την ε, τάξη σε όλες τους δήμους και κοινότητες. και εξασφαλίζουμε το σεβασμό των κανόνων. Υπάρχει διάλογος, εξασφαλίζουμε το διάλογο, ούτω ώστε να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία και ασκούμε και κάποια καθήκοντα, τα οποία ουσιαστικά είναι καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας. Με το διάταγμα 14 17 σε ό,τι αφορά τις, την ασφάλεια των πόλεων, ε, υπάρχουν δύο επίπεδα, ένα εθνικό και ένα τοπικό, ε, με βάση την αυτονομία των δημάρχων ε, και της τοπικής αστυνομίας ε, να ρυθμίζουμε την καθημερινή ζωή και την ασφάλεια στις πόλεις. Ε, όχι με αποκλειστικό τρόπο, αλλά ε, ακριβώς έχοντας τα ίδια καθήκοντα με την Εθνική Αστυνομία, συνεργαζόμενοι με την Εθνική Αστυνομία ε, στις παρεμβάσεις μας. Ε, κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών, είμαστε παρόντες σε τοπικό επίπεδο, και χρησιμοποιούμε όλα τα τεχνολογικά μέσα για να ελέγξουμε ε, τους, ε, τις περιοχές που κινδυνεύουν. Όλη αυτή την προσπάθεια την κάνουμε με βάση τον ε, ε, νόμο του 2018. κάνουμε, χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία όπως το Taser και τα λοιπά, ε, μπαίνουμε σε κτίρια, ε, κάνουμε μπλοκ στους δρόμους, ε, καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Ε, όλες αυτές τις δραστηριότητες τις ασκούμε εμείς με τη συνεργασία άλλων αστυνομικών. Επίσης, παρότι κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, υπαγόμαστε σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Νομίζω ότι αυτό είναι, γίνεται κατά παράβαση των κοινοτικών των δικαιωμάτων μας. Υπάρχει ένα διάταγμα ε, το οποίο ιδιωτικοποίησε την, την δημοτική αστυνομία, ενώ απέκλεισε τις υπόλοιπες αστυνομίες. Είμαστε λοιπόν θύματα διακριτικής ε, μεταχείρισης, γιατί ενώ ε, κάνουμε τα ίδια πράγματα, ε, δεν έχουμε, έχουμε διαφορετικές συμβάσεις. Μας ιδιωτικοποίησαν. Δεν είναι σωστό να μας ιδιωτικοποιήσουν. Αυτό είναι απαράδεκτη ε, διάκριση. Μιλάω τώρα για την δημοτική και επαρχιακή αστυνομία. Εμείς ασκούμε ε, δημόσια λειτουργία. Επίσης, ε, τα ωράριά μας που προβλέπονται και από τις ε, εθνικές διατάξεις και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ξεκάθαρα. Το άρθρο 2 του διατάγματος 93 ε, κάθετος 104 αφορά τα ωράρια των... που έχουμε εμείς. Ε, για όλους όσους ε, ασκούν αστυνομικές ε, δραστηριότητες και δουλεύουν σε σωσονιστικά ιδρύματα. όλα αυτά ισχύουν και η ενωσιακή νομοθεσία και η εθνική νομοθεσία ισχύει για τις υπόλοιπες αστυνομίες, αλλά όχι για μας. Ποια είναι τα δικαιώματά μας, ποια είναι η προστασία μας, τι εξασφαλίσεις έχουμε, τι σύμβαση έχουμε, τι προνόμια έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους της τοπικής αστυνομίας, ε, να φοράμε τη στολή, ε, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ε, πολιτών. Δεν κάνουμε πλάκα για την ασφάλεια των πολιτών. Ή είμαστε αστυνομικοί ή όχι. Το 2013 υποβλήθηκαν διάφορα ερωτηματικά στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για τους Αστυνομικούς Eurocop. Ε, επίσης, ε, ζητήσαμε και από την Ιταλική κυβέρνηση ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να, αναλύσουμε την παραβίαση του ευρωπαϊκού ε, εθιμικού δικαίου να μην σταματήσετε σε επιφανειακές απο, απαντήσεις της ε, Ιταλικής κυβέρνησης, να στείλετε επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση γιατί δεν πρέπει να πλένει ο σπόντιος Πιλάτος τα χέρια. Πρέπει να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκοί νόμοι, ε, γιατί εμείς συνεισφέρουμε στον έλεγχο της τρομοκρατίας, ε, ο οποίος δεν έχει σύνορα ούτε όρια. Ε, χρόνια προσπάθουμε να μιλήσουμε, συντό συγγνώμη που μακρηγόρω, ε, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στην Ιταλία. θα πρέπει ε, να λάβετε υπόψη σας ότι εμείς ε, προσπαθούμε, ερχόμαστε σε επαφή με επικίνδυνα άτομα, επικίνδυνα που τα ψάχνουμε ε, και είναι καταζητούμενοι επί χρόνια. συχνά δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε πληροφορίες. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ιταλία με διάφορους τρομοκράτες που κάνανε διάφορες απόπειρες και τρομοκρατικές ενέργειες με νεκρούς κτλ. Ε, εμείς ε, τι κάνουμε, εμείς παρεμβαίνουμε και ζητάμε στοιχεία του συχνά, ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους κινδύνους δηλαδή. Ε, και παρόλα αυτά τι σύμβαση έχουμε, μία ε, σύμβαση της ντροπή, ιδιωτικού δικαίου. Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι έχουμε θύματα κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Μα για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε πρέπει να σεβαστείτε το χρόνο σας. Αλλιώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. In order to discuss this thoroughly and... Για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό σε βάθος, οφείλετε και εσείς να σεβαστείτε το χρόνο που σας έθεσα. Να κλείσω. Τονίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρόεδρος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δράσεις για να έρθει σε επαφή ε, με την Ιταλική κυβέρνηση για να εξασφαλίσουμε η μεταχείριση στις συμβάσεις μας ανάμεσα στην ε, δημοτική και επαρχιακή αστυνομία και σε υπόλοιπε αστυνομικέ δυνάμει, για να υπάρχει καλύτερο έλεγχο στην Ιταλική επικράτεια και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για κοινο... τι κοινότητέ μα και για την Ευρώπη. Η τοπική αστυνομία είναι η αστυνομία που βρίσκεται επιτόπου στι κοινότητε. Ε... Βρίσκεται παντού. Κανένας δεν ξέρει τόσο καλά το, τους τόπους και τα άτομα που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι η μόνη η οποία μπορεί να ανακτήσει τις αξίες, την αρχή της ε, ε, εκπαίδευσης, το σεβασμό των άλλων ε, και την ανεκτικότητα απέναντι στου ανθρώπου μα. Ζητώ συγγνώμη που Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Σύντομη διόρθωση. Η αναφορά μας ήρθε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή όχι πριν από πολλά χρόνια, είναι του 2017. Άρα δεν ε, συνεχίζεται επί χρόνια και δεν κάνουμε πολύ τίποτα και άλλη μια διόρθωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες να παρέμβει. Αρμοδιότητα της Παρούσα επιτροπή είναι Αναφορών. Και αυτό προσπαθώ να βρω τώρα, δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο για να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημά σα. Προσωπικά θα μιλήσω με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ένας ε, αγαπημένο συνάδελφος και φίλος. Θα του θέσω το θέμα και θα τον ενημερώσω. Όμως ο ίδιο δεν μπορεί να ανατρέψει ό,τι κάνουμε εμεί εδώ στην παρούσα Επιτροπή Αναφορών. Άρα με εμά πρέπει να συνεργαστείτε. Να ακούσαμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Βαλεντίν ή ο κύριος Βάιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους αναφερομένους που προσήλθαν σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες για να αναπτύξουν το θέμα της αναφοράς των, κάτι που το οποίο μας βοήθη πολύ. Ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώνει τη συζήτηση αυτή και μας επιτρέπει έτσι να ακούσουμε τις ανησυχίες των άμεσα θυγωμένων. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σημαντικό ρόλο των αστυνομικών δυνάμεων και των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων στον αγώνα κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αστυνομικός, αλλά στην ομάδα την οποία, της οποίας ηγούμε αυτή ε, αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από αστυνομικού και τελωνιακού, από όλε τι χώρε μέλη. Κατανοώ και αντιλαμβάνομαι τη δυσχέρεια των καθηκόντων που ασκεί η αστυνομία και καμιά φορά υπό δυσχερεί συνθήκε και σε ένα ε, περιβάλλον μεταβαλλόμενο. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να εκφράσω την αναγνωρισή μου και να τονίσω ότι πληρώνει και βαρύ τίμημα. Πληρώνουν μάλλον και βαρύ τίμημα οι αστυνομικέ δυνάμει. Ε, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι και σημαντικό εργαλείο για να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των αστυνομικών δυνάμεων. Και εκεί οι τοπικέ αστυνομικέ δυνάμει παίζουν σημαντικό ρόλο. Η πρόληψη εγκλημάτων ασφαλώ και αποτελεί ε, αναπόσπαστο μέρο κάθε συνεκτική πολιτική και υπάρχει και πλατφόρμα χωρών μελών στην οποία ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη εγκληματικών δράσεων και ε, κάνουμε και μια εργαλειοθήκη για community policing, για ε, δημοτικές και κοινοτικές αστυνομίες. Η συνάδελφός μου, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελε και αυτή να πει λίγα λόγια για το δίκτυο αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, έχοντας πει αυτά ως εισαγωγή, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και ως θεματοφύλακα των συνθήκων οφείλουμε πρωτίστως να ακολουθούμε την συνθήκη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να επαναλάβουμε τα όσα είπαμε και παλαιότερα. Το άρθρο 72 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση λέει καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εντολή για να παρέμβει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών η τήρηση της εσωτερικής δημόσιας τάξης σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και συνεπώς είναι ζήτημα των χωρών μελών και εν προκειμένου της Ιταλίας να ρυθμίζουν τα των δυνάμεων ασφαλείας τους με τα όσα προβλέπονται στην εθνική τους νομοθεσία. Αυτό έχω να πω επί του παρόντος ε, και αν ε, επιτρέπετε από άποψη να μιλήσει και η συνάδελφός μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι και σημαντικός ε, ε, φορέας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται και σε ένα δίκτυο προσώπων που δρούν επί του πεδίου για να συλλέξει ε, σωστές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ριοπαστικοποίησης. Πρόκειται για δίκτυο που ε, αποτελείται από 10 ομάδες εργασίας και οι οποίες, ε, από τις οποίες ορισμένες αφιερώνουν τις προσπάθειές τους στην παρακολούθηση του έργου των αστυνομιών όλων των επιπέδων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού κλπ. Συναντώνται τρεις φορές το χρόνο ε, συζητούν και με άλλους φορείς. Όλοι μαζί λοιπόν ε, συμβάλλουν στην καθιέρωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για να βοηθήσουν όσους δρούν ε, στην πράξη για την αντιμετώπιση των ριζοσπαστικών απειλών κατά της ενωμιστάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Μου εξηγήσατε τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πω πολύ σύντομα. Ορισμένες φορές, σύμφωνα με τις συνθήκες, κάποια θέματα είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Όμω, έχουμε ενδιαφέρουσε εμπειρίε από την παρούσα Επιτροπή Αναφορών, διότι καμιά φορά χρειάζεται μια εξεταστική επίσκεψη, καμιά φορά χρειάζεται μια επιστολή, καμιά φορά μάλιστα χρειάστηκε απλώ να πάρω τηλέφωνο κάποιον υπουργό ή κάποιον δήμαρχο και αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Άρα, μην υποτιμάτε το έργο τη Επιτροπή μα. Τώρα, Ας ακούσουμε τους ε, συναδέλφους μας και πολύ ευχαριστώ να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσίριο. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Τσίριο. Πολύ σωστά αναδείξατε τη σημασία της Επιτροπής μας. Έχουμε αποσπάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, από επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ε, δηλαδή από συγκεκριμένα προβλήματα και πάρα πολύ σωστά οι αστυνομικοί εστράφησαν προς ε, εμάς και υπήρξε συνεννόηση με τον πρόεδρο Ταγιάννη και σίγουρα πρόκειται να υποστηρίξει τους τοπικούς κοινοτικούς τέλος πάντων αστυνομικούς της Ιταλίας που έχουν ιδιότυπο ρόλο Ε, φυσικά ο εγκληματίας δεν αλλάξει δηλαδή συμπεριφορά ανάλογα με τη στολή που βλέπει μπροστά του. Γιατί θα κάνει τη δουλειά του, είτε έχει μπροστά του καραμπινιέρο, είτε έχει την εθνική αστυνομία, είτε έχει την κοινοτική την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία τέλο πάντων. Οπότε και για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους θα πρέπει να βγουν από αυτή την τόσο παρά, παράλογη θέση. Έχω ασχοληθεί στο Πεδεμόντιο, στην περιφέρειά μου, κατά την πολιτική μου σταδιοδρομία με την αστυνομία και ξέρω ε, πώς, πόσο αξίζουν αυτοί οι αστυνομικοί. Είναι πολύ στριμωγμένοι επομένως και υπάρχει αυτή η επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών που μας έχει ε, διαβιβάσει φεβδοφέρα του 18 και εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. <laughs> τελικά συνομίλησε το Υπουργείο με τον αρχηγό τη Εθνική Αστυνομία. Ε, ναι, αλλά το συμφέρον τη Εθνική Αστυνομία δεν είναι να υποστηρίξει την τοπική αστυνομία. Βλέπουμε ε, την, ε, ε, την, απάντηση ότι είναι νομική, είναι τεχνοκρατική ούτω ή αυτή η απάντηση, δεν είναι πολιτική. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, Πρόεδρε, και οπότε γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να αποταθούμε στην κυβέρνηση, όχι στο Υπουργείο Ιστορικών που είναι απλώς ένα κομμάτι της κυβέρνησης. Οπότε και ο Πρωθυπουργό έχει την πολιτική ευθύνη να λάβει κάποιες αποφάσεις ούτω ώστε να αναγνωριστεί το λειτουργήμα ε, ε, που είναι κάτι, κάτι, κάτι γενικότερο, δεν είναι κάτι που αφορά συγκεκριμένα και μόνο το Υπουργείο Ιστορικών. Άρα να γράψουμε, να πούμε ότι πρόκειται για μια ανομαλία που είναι διαζώντως ε, Ιταλική. Γιατί έχουμε ε, τόση, αυτονομία, αλλά είναι παράλογο το ότι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή για τις σχέσεις της, ε, του, των δήμων, των πόλεων με ε, τους πόλεις δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί πρόκειται για συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχουν και για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα ε, ξεχνάμε. Δεν υπάρχει για τις συγκεκριμένε αρμοδιότητες της αστυνομία η τόσο ειδική οδηγία. Πάντως, γενικά οι οδηγίες δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε να εκμεταλλευτούμε την αρμοδιότητα που έχουμε να προσφύγουμε σε κάποια επίσημη καταγγελία, όπως γίνεται κάθε φορά που κάποιο κράτος δεν σέβεται το κοινωνικό δίκαιο. Χρειαζόμαστε πολιτική απάντηση, άρα να μας τα πει η Ιταλική κυβέρνηση. Δεν αρκεί αυτό το τεχνικό νομικό κείμενο του Υπουργείου Ιστορικών. Η Πρόεδρος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και Ξέρετε, δεν ζητούμε νομική απάντηση. Λογική, η κοινή λογική μπορεί να ισχύσει ακόμα και μέσα σε μια κυβέρνηση. Μιλούμε για προς κοινή λογική. Οι αστυνομικοί υπερασπίζονται τους πολίτες, τον κόσμο. Εάν αυτό καταρρεύσει, μα είναι απλό, είναι απλό ζήτημα κοινή λογική, εύκολο να λυθεί. Ο κύριος Μητροφάνος. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε λάβαμε την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Ότι δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσα θέματα έχουν σχέση με τη δημόσια ασφάλεια πρέπει να λύνονται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων των χωρών μελών. Όμως εδώ πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από την άποψη των διακρίσεων. Διάκριση δηλαδή ε, σε βάρος ενός μέρους εργαζομένων στο δημόσιο. Διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην κανονική αστυνομία και στην δημοτική αστυνομία. Έχασα κάποιες πληροφορίες από τις παρουσιάσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι των ε, αναφερομένων και <clears throat> υπάρχουν ορισμένα θέματα που ε, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό είναι ανοιχτό. Ποια είναι η θέση των συνδικάτων. Επιτρέπεται να δημιουργούνται να δημιουργούν οι αστυνομικοί συνδικάτα στην Ιταλία. Και ποια είναι η θέση της Ιταλικής Βουλής. Με ποια επιχειρήματα θεωρούν ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί στο επίπεδο της Ιταλικής Βουλής. Εάν το θέμα είναι μόνο οικονομικό, δημοσιονομικό, για να λυθεί δηλαδή το θέμα του καθεστώτος των ε, τοπικών αστυνομικών δυνάμεων. Είναι μόνο αυτό, είναι μόνο δημοσιονομικό ή πρέπει να αλλάξουν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις. Και το άλλο είναι το θέμα πώς χρηματοδοτούνται οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις από τους προϋπολογισμούς των κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων δηλαδή, ή από τον κεντρικό προϋπολογισμό του Ιταλικού κράτους. Και τι θα συμβεί εάν οι τοπικοί αστυνομικοί αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι κανονικοί αστυνομικοί. Μπορεί να πει κανείς ότι θα είναι καλύτερα προστατευμένοι. Όμως δεν γνωρίζουμε ποιες νέες υποχρώσεις θα κληθούν να αναλάβουν. Και τι είδους καθήκοντα θα πρέπει να ασκούν εφόσον έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα και υποχρώσεις με τους κανονικούς αστυνομικούς. Το συμπέρασμά μου είναι το εξής. Να συνεχίσουμε την διαρεύνηση της ε, αναφοράς αν είναι δυνατόν να γράψουμε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας και στην Ιταλική Βουλή και να ρωτήσουμε εάν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα αυτό ενδεχομένω και ενώπιον του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ίσως είναι δηλαδή δυνατόν να γίνει αυτό υπό την έννοια της ε, αποφυγής διακρίσεων. Υποστηρίζουμε η ομάδα μου δηλαδή και εγώ την αναφορά των Ιταλών τοπικών αστυνομικών και τον αγώνα που κάνουν για την εξασφάλιση των δικαίων τους. Ευχαριστώ πολύ. Ελεονόρα Εύη, είμαι βεβαία ότι εσείς θα είστε συντομοτάτοι και ότι ε, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως πάντα Πρόεδρε προσπαθώ να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους ε, αναφέροντας που ξανακατέβασαν την ε, αναφορά τους. Μας την ξαναεπέβαλαν, ούτω ώστε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα το οποίο τραβάει εδώ και πολύ καιρό. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συναδελφοί, είναι τρομερή αυτή η δυσμενής διάκριση. Δεν δικαιολογείται, είναι παράλογη. Θα πρέπει το θέμα να επιληθεί όσο γίνεται συντομότερα. Και είδαμε, ε, κάνουν τόσα πράγματα που κάνουν και άλλες αστυνομίε, Γιατί να έχουν εγγυήσει διαφορετικές υπέρ αυτών και θέλω να σας ε, υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει κάποιες ε, απόπειρε και κατά αυτή την ε, θητεία και κατά αυτή τη θητεία της κυβέρνησης των πέντε αστέρων προσπάθειες για να λιανθούν αυτές οι διαφορές. Οπότε και σήμερα η κυβέρνησή μας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας που έχουμε παρουσιάσει στο λαό της χώρας, προσπαθούμε να λύσουμε και αυτά τα προβλήματα της τοπικής αστυνομίας. Γιατί, είπαμε, κρεμούν πολύ καιρό. Λίγα έχουν γίνει Έχουμε ένα μικρό βήμα με ένα διάταγμα για την ασφάλεια και έτσι εν μέρη κάτι κάνουμε για το πρόβλημα. Για την τράπεζα δεδομένων, για την πρόσβαση από τους αστυνομικούς, για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά σίγουρα αυτό δεν αρκεί θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θα πρέπει να αποκλειστούν όσες δυσμενείς διακρίσεις ακόμα από Να ισχύουν τα ίδια όπως και με τις άλλες αστυνομίες. Σχολείο με την ασφάλεια και εμείς θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ως πολίτες για το έργο που επιτελεί η τοπική αστυνομία και συμφωνώ με τους συναδέλφους να απευθύνουμε αυτή την επιστολή στο Υπουργείο Ιστορικών να εξετάσουν με τόλμη με σοβαρότητα το θέμα για να λυθεί το μητώδιο. Συνομοτρουδινάτων ευχαριστούμε τους αναφέροντες και πάλι. Η Πρόεδρος Γιάρ. Ευχαριστώ. Με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Με τη ζωική πορεία των πραγμάτων. Θα πρέπει κανείς να έχει μια λογική προσέγγιση. Και θα πρέπει να βοηθήσουν και οι τοπικές αρχές να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Να το πούμε αυτό στην επιστολή μας. Αυτό να είναι καλή αφετηρία. Να ξεκαθαρίσουμε στην επιστολή μας. Ότι μας προβλήζει πάρα πολύ. Ότι δεν έγινε τίποτε από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή αυτή τη αναφορά. Σε λίγο ολοκληρώνεται αυτή η θητεία αλλά θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πρέπει να γίνει και κάποιο είδου ε, αποστολή εξακρίβωση των πραγμάτων στην επόμενη θητεία και να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι που τίποτα δεν έχει γίνει και αυτό σημαίνει δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Πίτερ, σε ευχαριστώ και εγώ νομίζω ότι μια ερευνητική αποστολή θα ε, ήταν χρήσιμη. Είπαμε ότι η αποστολή του Υπουργείου ήρθε το Φεβρουάριο του 2018 και τι θα γίνει. Έχουμε άλλωστε και τι εκλογέ. Κυρία Τόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ τους αστυνομικούς και τις ενώσεις τους και τα μέλη της τοπικής αστυνομίας που ήρθαν εδώ για δεύτερη φορά. Σας ευχαριστώ γιατί έχετε συνέπεια. Αποδείξατε ότι δεν θα σταματήσετε για να δικαιωθείτε. Αυτό που ζητάτε είναι σωστό. Ε, και φαίνεται ότι έχετε εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στην Επιτροπή μας και στην Πρόεδρό μας. Ε, ακριβώς αυτή η εμπιστοσύνη μας δεσμεύει και εμάς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά τους με ανάλογη σοβαρότητα. Σας είπαμε ότι το Φεβρουάριο ε, στείλαμε την... Ε, επιστολή. Το Μάρτιο έγιναν οι Ιταλικές εκλογές. Ε, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Η κυρία Εύη μίλησε για αυτή. Εγώ εκπροσωπώ την, α, τους σοσιαλιστές και δημοκρατικούς και σας στηρίζουμε σε αυτή τη μάχη. Ο πρώτος ε, παραλήπτης της επιστολής ε, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Ε, είναι αρμόδιος όχι μόνο για την αστυνομία, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, και επειδή η τοπική αστυνομία ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ε, πραγματικά ανήκει στο χαρτοφυλακιό του. Δεύτερον, υπάρχει και ολόκληρη κυβέρνηση. Πρέπει να γράψουμε σε ολόκληρη την κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να στείλουμε και στον πρόεδρο Φίγκο και στον ε, πρόεδρο Καζελάτη στην, ε, στο κοινοβούλιο, δηλαδή στο Ιταλικό κοινοβούλιο, στα δύο σώματα της Βουλής, ε, μια επιστολή. Για να κάνουμε λοιπόν τα πάντα, να καλύψουμε τους πάντες, να σας πω ότι μας δώσαστε σαφείς απαντήσεις, αλλά προφανή πράγματα μας είπατε. Μας είπατε ότι ασχολείστε με την ασφάλεια. Ε, ξέρουμε ότι εκπαιδεύεστε κι εσείς, αλλά σας ζητάμε κάτι παραπάνω. Ε, θα πρέπει να μας βοηθήσετε για να βρούμε την κατάλληλη νομική βάση για να μπορέσει και η Κομισιόν να κάνει ό,τι πρέπει απέναντι στο Ιταλικό κράτος. Τέλος, η αποστολή. Συμφωνώ με την Πρόεδρο, χρειάζεται να γίνει μια αποστολή στην Ιταλία και εμεί είμαστε στην τελική φάση τη κοινοβουλευτική θητεία. Αν έχουμε το χρόνο και τι προποθέσει, νομίζω ότι θα μπορούσε μια ομάδα ευρωβουλευτών να πάει επί τόπου και να πιέσει ε, με αποφασιστικότητα για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα συμμεριζόμαστε απόλυτα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thanks to you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε ε, για το γεγονός ότι υπάρχουν 60.000 δημοτική αστυνομική, τοπική αστυνομική στην Ευρώπη που αντιμετωπίζονται με άδικο τρόπο, θύματα διακρίσεων. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την επιστολή, την αναφορά, να στείλουμε ε, μία ναι μεν ευγενή αλλά ειλικρινή επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση ε, και αντίγραφο στην ε, Ιταλική Βουλή. Γιατί μιλάμε για εκλεγμένους εκπροσώπους που ασχολούνται με θέματα εσωτερικών ε, και κοινωνικών υποθέσεων της χώρας τους, πρέπει να τους στείλουμε και αυτόν την επιστολή. Επίσης, πιθανή ε, αποστολή στην Ιταλία που θα γίνει όμως με το νέο κοινοβούλιο, θα το αποφασίσει η νέα Επιτροπή Αναφορών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι ένα από αυτά που είπατε. Να αποδείξουμε ότι είναι μία δουλειά και μία αποστολή, ανεξάρτητα από το, την ονομασία του, της αστυνομίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική και ενιαία προσέγγιση απέναντι στα αστυνομικά σώματα. Πιστεύω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει πάντα ο τρόπος να προχωρήσει κανείς και να βρει λύση. Αυτό που θέλω να κάνω με αυτή την επιστολή είναι να κινητοποιήσω την Ιταλική κυβέρνηση για να μπορέσει το συντομότερο δυνατόν να αποκαταστήσει τα δικαιώματα αυτών των 60.000 δημοτικών και επαρχιακών αστυνομικών δηλαδή τοπικών αστυνομικών που αντιμετωπίζονται άδικα, ε, υφίστανται διακρίσεις και να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τους εθνικούς αστυνομικού. Ακριβώ αυτό πρέπει να κάνουμε, να κινητοποιήσουμε την ε, κυβέρνηση και να τους δείξουμε πόσο άδικο είναι αυτό για να προχωρήσει, να κάνει κάτι. Αυτό νομίζω μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή τη φάση. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά στον Αντώνιο Ταγιάννη για το θέμα αυτό. Ε, είμαι σίγουρη ότι παρακολουθεί εκ σε αυτό το θέμα, γιατί μια ε, έτσι παρατυπία, ας πούμε, πρέπει να διορθωθεί. Συμφωνούν οι συνάδελφοι μαζί μου. Σούπερ, πολύ ωραία. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την αποστολή, για αυτή την αναφορά, συγγνώμη. Ε, και σας ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να έρθετε στις Βρυξέλλες. Εγώ βλέπω κάτι που δεν βλέπετε. Χιονίζει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. I'm sure that it has been a sacrifice by you to... Θυσιάσατε πολλά. Φύγατε, φύγατε από την όμορφη Ιταλία για να έρθετε σε αυτή την πολύ ζωφερή εικόνα της, ε, γωνιά της Ευρώπης, για να δείτε αυτή την θλιβερή εικόνα. Ε, καλό ταξίδι στην ε, στη Μεσόγειο. Στην Ιλιόλου, στη Μεσογειακή σας χώρα. Thank you so much and I believe that you are now leaving us. Τώρα ήρθε η ώρα να μας αφήσετε. Ας κάνουμε ένα μονόλεπτο διάλειμμα μέχρι να φύγετε και κατόπιν θα αρχίσουμε να συζητούμε την επόμενη αναφορά. Η Πρόεδρος, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ προσέξτε, προσέξτε το επόμενο θέμα, το οποίο αφορά διπλή τιμολόγηση για ηλεκτρικό και νερό. Έχουμε τους ε, αναφέροντες εδώ, που είναι η Πατρίσια Γκρέαμ. Πέντε λεπτά έχετε για να παρουσιάσετε την αναφορά σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα. Να σας πούμε τι γίνεται με αυτές τις κοινόχρηστες υπηρεσίες. Έχουμε δύο ταρίφες. Πρώτα-πρώτα για τους μόνιμους κατοίκους και άλλη τιμή για τους μη μόνιμους κατοίκους είναι πιο φτηνό για αυτούς που έχουν εκεί την ε, κυρία τους κατοικία. Επίσης, για αυτούς που έχουν δευτερεύουσα ε, κατοικία, πληρώνουν περισσότερα από όσο αυτοί που είναι με κάτοικοι. Και ε, θέλω να σας πω ότι αυτοί, αυτές οι τιμές ε, δεν επιβάλλονται αυτοδίκαια. Θα πρέπει κανείς να καταλάβει τι ισχύει. Ισχύει για την κυρία κατοικία κάποιου προσώπου, αλλά σας τονίζω ότι θα πρέπει κανείς να κάνει ε, αίτηση. Δεν ε, χορηγείται αυτοδικαίως. Η άλλη πιο ακριβή τιμή, ε, εάν δεν γίνει αίτηση, ισχύει για όλους. Αν δεν γίνει αίτηση για το χαμηλότερο τιμολόγιο. Οπότε, αν κανείς δεν ξέρει τι προβλέπεται για τη διαφορετική τιμολόγηση, τότε αυτομάτως πληρώνουν στα περισσότερα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για μια οικογένεια έξι προσώπων θα ήταν 99,77 το μήνα και ακριβώς για την ίδια κατανάλωση, αλλά για την πιο ακριβή ταρίβα δεν είναι 155,29. Είναι τερατώδης αυτή η διαφορά. 63,52 τον ε, μήνα. Οπότε το χρόνο αυτό σημαίνει 762 ευρώ. Και είμαι σίγουρη ότι θεωρείται ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος για την μέση οικογένεια. Οι περισσότεροι φρικιούν όταν συνειδητοποιούν πόσο παραπάνω πρέπει να πληρώσουν. Και ε, πολλές φορές ο σπιτονικοκύρης που νοικιάζει ή ε, το η κυβέρνηση για τις εργατικές κατοικίες ε, σε σχέση με την ε, εταιρεία υδάτων θα πρέπει για τις δέκονε ενημερωθούν για να δουν πώς θα ενημερώσουν μέσω κάποιου website αλλά πού να το ξέρει όποιος έρχεται στη χώρα δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αυτή την τόσο σημαντική διαφορά στην τιμολόγηση. Δεν έχουν δικαιώματα οι ενοικιαστές. Αυτό είναι υπερβολικό. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ε, ό,τι θέλει κανένας κάνει στην αγορά των εκμισθώσεων. Δεν υπάρχει προστασία για το μισθωτή έναντι τέτοιων πρακτικών. Οι πάρα πολλοί μισθωτές ποτέ δεν βλέπουν καν τον ε, λογαριασμό. Πληρώνουμε το νίκη ένα σταθερό ποσό και πολλές φορές αυτό το ποσό δεν έχει καμία σχέση με το τι λέει ο μέτρητής. Οι μισθωτές που καταλαβαίνουν τι γίνεται πάνε και βρίσκουν τον σπιτινικό κύριο και ζητούν να υπάρχει στον λογαριασμό ρητή ανάλυση. Ε, ε, πολλές φορές όμως λέει ο εκμισθωτής όχι. εμεί γι' αυτό κάνουμε και την αναφορά Θέλουμε με την αναφορά όλοι να πληρώνουν το, το ίδιο για, τον, για το, το, ηλεκτρικό ακριβώς πως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αφού έχουμε ένα τέτοιο σύστημα διπλής τιμολόγησης ε, το οποίο είναι νόμιμο γιατί να μην γίνεται αυτό και σε άλλες χώρες και πολλοί εκμισθωτές δεν το κρύβουν ότι φοροδιαφεύγουν και εάν δεν υπάρχει σχετική διαδικασία τότε θα ψήφι... αν κάνει τη σωστή διαδικασία ο, ο μισθωτής τότε θα ξαναδόν το ο φόρος θα πληρώσει ο εκμισθωτής και γι' αυτό το λόγο πολλοί δεν θέλουν την μισθωτική σύμβαση και φεύγουν από εκεί που μένουν και πηγαίνουν για να βρουν φθηνότερες τιμές κάπου αλλού. Όμως, αν καταγγείλουν την ε, σύμβαση οι μισθωτές, τότε ο εκμισθωτής θεωρεί ότι αυτό είναι παράνομο και τότε δικαιούνται την εγγύηση που έχει καταβάλει ο μισθωτής στην αρχή της ε, σύμβασης. Άρα Έτσι ο μισθωτής δυσκολεύεται να έχει τη φθηνότερη τιμή. Ναι, αλλά και υπάρχει και το έντυπο H για να μπορεί να ωφεληθεί από την φθηνότερη τιμή. Τώρα θα πρέπει να κάνει μια έτσι με 50 ευρώ για να φτάσει στα 466. Ακόμα χειρότερα. 13% είναι η τιμή για την διόρθωση κάποιων ε, σφάλματων και ακόμα χειρότερα. Άλλα 50 ευρώ για ε, διοικητικά έξοδα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, λέει πρόεδρος, γιατί έχετε υπερβεί το συγκεκριμένο χρόνο που σας διατίθεται. Επίσης, οι τυχεροί που έχουν κάποιον σπιτονικό κύριο που κάνει το, το, σωστό και που συμπεριφέρεται με τρόπο υπεύθυνο, ε, τότε τους καταχωρεί και αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιο είδου χρέωση, κάποια επιβάρυνση για αυτούς τους ενοικιαστές. Ή πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ε, εκπροσωπείται εδώ, Παρακαλείται να ε, εξηγήσει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν πράγματι διαφορετικά τιμολόγια στην Μάλτα. Και όσο εξηγήθηκε στην αρχή, δεν υπάρχει πρόσβαση στο μειωμένο τιμολόγιο για Ευρωπαίους πολίτες. Έχει προχωρήσει σε ε, προσφυγή για παραβίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Μαλτέζικες αρχές ε, ε, υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν και τα ποσά τα οποία έχουν αχρεωστεί τους καταβληθεί. Ε, πράγματι, η κατάσταση τώρα ε, προβλέπει ότι ο, ο μπορεί να υπογράψει το έντυπο H και ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει με το έντυπο F το μειωμένο τιμολόγιο. Αλλά πρέπει να κάνει μια κατάθεση, να καταθέσει ένα ποσό πρώτα. δεν υπάρχει διάκριση πλέον μεταξύ Μαλτέζων πολιτών και πολιτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι μισθωτές ανεξαρτήτως εθνικότητας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μειωμένο τιμολόγιο. Η μόνη διαφορά λοιπόν που μένει πλέον είναι ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον μισθωτή. Ο μισθωτής καλείται να καταβάλει την παρακαταθήκη αυτή για την διασφάλιση δηλαδή του ότι θα πληρώνει. Εάν δηλαδή ο μισθωτής δεν πληρώνει τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, θα είναι και δύσκολο να, μάλλον θα μπορεί ο εκμισθωτής να πάρει τα χρήματα που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια. Ευχαριστώ. Α, εσείς, ποιο είναι το όνομα, πώς είναι το όνομά σας. Α, Κατούριο από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για θέμα το οποίο άπτεται και τη νομοθεσία για προστασία καταναλωτών, αλλά και την ε, νομοθεσία περί ενέργειας. Ακούσαμε την άποψη των καταναλωτών, ας ακούσουμε τώρα και την νομοθεσία για την ενέργεια. Ένα από τα μεγάλα θέματα εδώ είναι γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά τιμολόγια και γιατί είναι νόμιμο αφού δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα μέλος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ρυθμιζόμενα τιμολόγια, δηλαδή τιμολόγια όπου η χώρα μέλος ρυθμίζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προβλέπεται, επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμως η... Μάλλον δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμως η Μάλτα έχει εξαίρεση, δηλαδή μπορεί να ρυθμίζει τις τιμέ των τιμολογίων όπως θέλει και για λόγους προστασίας καταναλωτών, διότι της Μάλτα είναι πολύ μικρό και απομονωμένο σύστημα. Εκεί λοιπόν είναι καλύτερα η κυβέρνηση να θεσπίζει τις ε, ε, τιμές αντί για κάποιο μονοπόλιο. Προτίμησε η Μάλτα λοιπόν το διπλό τιμολόγιο, όπου το οικιακό τιμολόγιο είναι κάτω του κόστους, δηλαδή επιδοτείται, είναι επιδοτούμενο τιμολόγιο και το νορμάλ ε, τιμολόγιο είναι σύμφωνο, ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος. Όπως είπα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αυτό είναι απόλυτα νόμιμο για τον απλό λόγο ότι η Μάλτα διαθέτει εξαίρεση από την ε, νομοθεσία της οδηγίας περί ηλεκτρικού ρεύματος. Το άλλο θέμα που αναφέρθηκε πριν εδώ είναι ως ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας που δεν είναι ιδιοκτήτης να αποκτήσει το τιμολόγιο αυτό. Και αυτό είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Ενέργειας, δηλαδή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και ο μισθωτής να ε, ε, έχει σύμβαση με την, με την παροχής ηλεκτρικού ρεύματο. Όποιο έχει λοιπόν λογαριασμό για πάνω από τρει μήνες μπορεί να λάβει το τιμολόγιο αυτό. Από καθαρά νομική άποψη λοιπόν είναι, έχουν καλώ τα πράγματα στη Μάλτα. Τουλάχιστον ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί ενέργειας. Πρώτο λοιπόν είναι υπάρχει, δεύτερο μπορεί να εφαρμόζεται. Δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει αυτό που του επιτρέπει ο εθνικός νόμος. Εδώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη σχέση μεταξύ του πελάτη ε, και, του παρόχου. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όμως έχει προβλέψει ένα μηχανισμό επιλύσεως διαφορών ακριβώς για να επιλύονται τέτοια θέματα. Εάν ένας πελάτης, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να έχει το οικιακό τιμολόγιο δεν το λαμβάνει, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στον μηχανισμό επιλύσεως διαφορών που χειρίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη Μάλτα και εδώ είναι το θέμα. Αν έχετε στοιχεία ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών δεν λειτουργεί σωστά, τον ρόλο δηλαδή που το έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τότε εμείς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο και να την κυνηγήσουμε τη Μάλτα, διότι η ρυθμιστική αρχή της δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Όμως η διαδικασία είναι ότι ο καταναλωτής πρέπει πρώτα να αποταθεί στον, ε, στη ρυθμιστική αρχή για τον μηχανισμό επιλύσεως διαφορών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνησή σας πραγματικά, ε, ακριβέστατη. Ας ε, δούμε τώρα τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Η Μαλτέζα, συνάδελφό μας, συνάδελφός μας Ροπέρτα, ήρθε πραγματικά ακριβώς ε, στο, χρόνο. να με συγχωρείτε, έκανα μια εγγραφή για την ε, τηλεόραση. Δεν θέλω να απόσχω από τα είπε ο, ο, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονό όμω ότι η αναφερομένη η κυρία Γκραμ αλλά και άλλοι ε, είναι εδώ παρούσα δείχνει ότι το θέμα δεν έχει επιληθεί. Είναι άρα ζήτημα ε, εντιμότητας, δικαιοσύνης και κάτι το οποίο αναμένει κανεί για κάθε πολιτική και ιδίω όταν έχουμε απέναντί μα ανθρώπου που είναι ε, υπήκοοι χωρών μελών. Παραμένουν θέματα ανοιχτά, εκκρεμεί. Πόσοι μισθωτές χρησιμοποίησαν το έντυπο F2 για ε, την αναγνώρισή τους ως ε, ε, μισθωτών που έχουν δικαίωμα να έχουν το οικιακό τιμολόγιο και πόσοι από αυτούς επέτυχαν να λυθεί το θέμα τους. Επίσης, πόσες ε, κατοικίες στη Μάλτα, ε, θερινές κατοικίες δηλαδή, ε, έχουν υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού κλπ. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Και δεν είμαι βέβαια ότι οποιοδήποτε μηχανισμό επιλύσεω διαφορών ή άλλη ρυθμιστική αρχή έχουν όντω αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχιστεί η συζήτηση και να μην δεχθούμε απλώ ότι κλείνει η παρούσα αναφορά. Άλλο κανεί παρακαλώ λέει η πρόεδρο. Καλώ. Επανέρχομαι στην αναφερομένη. Αλλά πραγματικά πολύ σύντομη παρέμβαση αυτή τη φορά. Έχετε ένα λεπτό. «466 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Για οποιονδήποτε στη Μάλτα να τα πληρώσει, μόνο και μόνο για να πάρει κάτι που δικαιούται. Και όπως είπε και η Ρομπέρτα, πρέπει να το επιλύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί το F2 δεν είναι ε, προσβάσιμο από ανθρώπους που παίρνουν το βασικό μισθό στη Μάλτα. Κλείνει το μικρόφωνο. Ε, ε, πρόκειται για πολλά χρήματα. Είναι σχεδόν τρεις μήνες ε, μισθού ενός μέσου προσώπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Είναι σημαντικό όντως να επιληθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ένα κατεπίγοντα χαρακτήρα. Θα κάνουμε το εξή. Διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά και επειδή έχουμε ήδη απευθυνθεί στις 17 Δεκεμβρίου στην κυβέρνηση της Μάλτας, δηλαδή πριν από ένα μήνα και ακόμη αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης ε, της Μάλτας. Ζητήσαμε δηλαδή στην επιστολή μας αυτή οι πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες αυτές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ε, δικαστηριών στην Μάλτα. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την απάντηση και στην ε, ε, διάρκεια αυτή θα κρατήσω με ανοιχτή την αναφορά. Ήταν άλλωστε ενδιαφέρον τουλάχιστον για μένα να δω ότι ο μηχανισμός επιχειρήσεως διαφορών που είναι άλλωστε υποχρεωτικός στις χώρες μέλη. Δεν ξέρω αν τον χρησιμοποιούν ή όχι ενδιαφερόμενοι. Εάν όχι τότε αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά για την ώρα σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ ενώπιόν μας, που φωτίσατε την υπόθεση και το γεγονός ότι συνεχίζουν τα πράγματα αυτά Ας περιμένουμε την απάντηση τη μαλτέζικης ε, κυβέρνησης και όταν θα λάβουμε την απάντηση αυτή θα δούμε τι είδους δράση θα λάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και, α, βλέπω ότι ακόμα χιονίζει στι Βρυξέλλες, βεβαίω, όχι στην Μάλτα. Ε, να επιστρέψετε λοιπόν στην όμορφη ε, νήσο σας ε, με ασφάλεια. Ας έλθουμε τώρα στην παρουσίαση μελέτης με θέμα διαφορές ποιότητας στα καταναλωτικά προϊόντα πολύ ευχαρίστως να δώσω τον λόγο στην Μπλάνκα Βίτοβα. Where do we have our expert? Έχει έρθει ο εμπειρογνώμονας. Α, έρχεται. The floor is yours. Thank you very much. Έχετε το λόγο λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχετε ακούσει για το θέμα της διπλής ποιότητας προϊόντων στην ενωσιακή αγορά, στην ενιαία αγορά. Ήρθα εδώ να κάνω μια νομική ανάλυση για τον κανονισμό ε, για τη διτή ποιότητα ε, των ίδιων προϊόντων ε, όπως προτείνεται το 2018. Ε, ή μάλλον, ε, όχι διπλή ποιότητα, όσο διπλή σύνθεση. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια αρχικά ήταν μια, αρχική, μια μεμονωμένη πρωτοβουλία κάποιων ευρωβουλευτών και εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με αυτό το θέμα συνολικά. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά τη. Η διτή ποιότητα. Ε, με την ίδια όμως επισήμανση ε, για τα προϊόντα σε διαφορετικά κράτη-μέλη έχει να κάνει κυρίως με τρόφιμα, ε, αλλά και ε, είδη ε, τουαλέτας, ε, καθαριστικά, καλλιντικά κτλ. Ε, πρόσφατα έχουμε κάνει ανάλυση του, του περιεχομένου σε εγκεκριμένα εργαστηρία σε κάποιες χώρες, στη Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Σλοβακία. Η ποιότητα προϊόντων Πώ αντικατοπτρίζεται στον ε, έμπορο. Καταρχά βάζει ε, προϊόντα με διάφορη σύνθεση, βάρος, ε, ποιότητα ή γεύση, αλλά με την ίδια συσκευασία, χωρίς να καταλαβαίνει σαφώ ο κατανολωτή και πέραν πάση αμφιβολίας για το γεγονό αυτό, για το ότι είναι δηλαδή άλλο προϊόν, με άλλο βάρος, άλλη σύνθεση κτλ. Η διπλή ποιότητα Μπορεί όμως να συμβαίνει όταν ο έμπορος βάζει ένα νέο προϊόν σε μια νέα αγορά και χρησιμοποιεί ένα προϊόν με καλύτερη σύνθεση, όπως υψηλότερο ποσοστό, υψηλότερη ποιότητα ε, κρέατος στη σύνθεσή του, ε, ε, εφιστά την προσοχή του καταναλωτή σε αυτή την υψηλότερη ποιότητα και μετά από κάποιο χρόνο το αρχικό προϊόν αποσύρεται από αυτή την αγορά και αντικαθίσταται από ένα προϊόν το οποίο είναι αλλοιωμένο, χειρότερη σύνθεση, αλλά με την ίδια μορφή, με την ίδια όψη. Ο καταναλωτή είναι πεπισμένο ότι αγοράζει το ίδιο προϊόν, γιατί δεν ε, έχει δει ποια είναι η σύνθεση του προϊόντος και δεν τσεκάρει τα συστατικά κάθε φορά που αγοράζει το προϊόν εφόσον έχει την ίδια συσκευασία. Ακόμα και αν ήθελε να ελέγξει τη σύνθεση, δεν θα θυμόταν ποια ήταν η σύνθεση του αρχικού προϊόντος, άρα με τι να το συγκρίνει, με τι να συγκρίνει το νέο προϊόν. Αυτό είναι η βαθμιαία ε, υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Με τη διπλή ποιότητα ε, τα προϊόντα περιέχουν τις ε, υποχρεωτικές πληροφορίες που προβλέπει η νομοθεσία ρητά σε κάποιες περιπτώσεις, σε περίπτωση ας πούμε, τροφίμων. Αυτές οι πληροφορίες Όμω έρχονται σε σύγκρουση με τη συνολική ε, εμφάνιση του προϊόντο, όψη του προϊόντο. Σε περίπτωση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών που αναφέρονται συχνά ε, στα προβλήματα διπλής ποιότητας, η αντίληψη του, η εντύπωση του καταναλωτή παίζει σημαντικό ρόλο. Σε περίπτωση τέτοιων προϊόντων διπλή ποιότητα, μπορούμε να πούμε ότι ο μέσο καταναλωτή κρατάει μόνο ε, συγκεκριμένε πληροφορίε. Ε, και δεν ε, διαβάζει και τις ε, τελευταίες λεπτομέρειες, ας πούμε. Ξέρει απλώς τη γενική όψη. Ε, κυρίως ε, έχει μια εικόνα για το προϊόν, αυτό του εντυπώνεται και επηρεάζει κυρίως την απόφασή του για το αν θα αγοράσει το προϊόν ή όχι. Αυτή η αντίληψη που έχει, η εικόνα που έχει για το προϊόν. Υπάρχουν διάφορα νομικά μέτρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την διπλή ποιότητα των προϊόντων. Και από το κανονισμό για το δημόσιο δίκαιο και το ιδιωτικό δίκαιο. Ε, ελαττωματικές επιδόσεις, ε, προβλήματα στον, ε, στη σύμβαση, προβλήματα με το δίκαιο ανταγωνισμού ε, και το δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οδηγία για τις αθέντες εμπορικές πρακτικές και με μονομένες συστάσεις κανόνες στον τομέα των, των ή ε, τροφίμων. Δεν λύνουμε όμως ε, επιτυχώς το πρόβλημα αυτό ε, των προϊόντων διπλής ποιότητας. Να εστιάσω στα πιο συγκεκριμένα μέτρα. Στη χρήση της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Η οδηγία αυτή θέλει να εμποδίσει πρακτικές του επιχειρηματία που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή και μπορεί να επηρεάσουν τον καταναλωτή στις διαδικασίες που θα κινήσει. Ε, αυτά αφορούν όλες τις τάσεις ε, της, ε, τις συμβατικές. Δηλαδή στην προσυμβατική φάση, όταν διαπραγματευόμαστε και συνάπτουμε την σύμβαση, αλλά ακόμα και μετά την, την υλοποίηση των υποχρεώσεων του επιχειρηματία. Τα διοικητικά σώματα θα κάνουν ένα, μια δοκιμή για τις αθέμητες πρακτικές ε, ενδεχομένως του επιχειρηματία. Στην πρώτη δοκιμή, στην πρώτη φάση, πρέπει να αξιολογήσουμε εάν οι εμπορικές πρακτικές πληρούν τα κριτήρια κάποιων από τις λεγόμενες αθέμητες εμπορικές πρακτικές που αναφέρονται στο μαυροπίνακα του πράγματο 1 τη οδηγία. Εάν η πρακτική δεν ε, καλύπτεται από τα κριτήρια του μαυροπίνακα, ε, τότε κάνουμε το δεύτερο τεστ. Αξιολογούμε αν οι πρακτικέ ε, πληρούν τα κριτήρια επιθετικών εμπορικών πρακτικών. Εάν τα κριτήρια των επιθετικών εμπορικών πρακτικών δεν πληρούνται, τότε εξετάζουμε αν η συμπεριφορά, η δράση, η παράληψη δεν πληρεί τα κριτήρια των παραπλανητικών εμπορικών εμπορικών πρακτικών με βάση το άρθρο 6 ή 7 της οδηγίας. Τέλος, εάν το διοικητικός, ε, ο διοικητικός φορέας λέει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν παραπλανητικές πρακτικές μπορούμε να αξιολογήσουμε αν η συμπεριφορά ε, μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικά αθέμητη εμπορική πρακτική. Ε, εάν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, η πρακτική δεν είναι αθέμητη. Ο κανονισμός για τις ε, παραπλανητικές ε, εμπορικές πρακτικές δεν αναφέρεται ρητά στη διτή ποιότητα, διπλή ποιότητα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ετοίμασε μια πρόταση με βάση ε, τις οποίες θα, της οποίας θα τροποποιηθεί η σχετική οδηγία. Θα υπάρχει παραπλάνηση αν υπάρχει θέση στην αγορά ενός προϊόντος ε, το οποίο λέγεται ότι είναι ίδιο με προϊόν που κυκλοφορεί σε άλλες χώρες, ενώ έχει τελείως διαφορετική, ουσιαστικά διαφορετική σύνθεση ή ε, ή χαρακτηριστικά, τα γενικά κριτήρια για να αξιολογήσουμε την ε, παραβίαση αυτής της ε, διάταξης που βλέπετε, συνοψίζεται ως εξή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά της πρακτικής θα πρέπει να προκαλεί ε, την, να, επηρεάζει την απόφαση του μέσου καταναλωτή και και ο καταναλωτή παίρνει ε, την απόφαση να προβεί σε μία συναλλαγή που δεν θα έπαιρνε διαφορετικά. Ε, δεν θα έπαιρνε σε διαφορετική προήπτωση. Ε, θα πρέπει να θα πρέπει το προϊόν αυτό να υπάρχει σε διάφορα κράτη-μέλη και σε κάθε κράτος μέλος να έχει διαφορετική σύνθεση, ουσιαστικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει τώρα να γίνει μια μεγαλύτερη ανάλυση και επειδή δεν έχω χρόνο θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο προβληματικά κριτήρια στην σημαντικά διαφορετική σύνθεση και σε επιπλέον κριτήρια βοηθητικά που αναφέρονται στο προήμιο της πρότασης. Το κριτήριο της σημαντικής διαφοράς θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε επιμέρους περίπτωση. Όταν αξιολογούμε την σημασία της διαφοράς, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιεί, ε, το ιδιωτικό δίκαιο σε περίπτωση ε, λάθους στη συμπεριφορά, ουσιαστικά διαφορές ε, στη σύμβαση ή παράβαση μιας σύμβασης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια σημαντική διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι ένα άτομο που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση θεωρεί ε, κάποια χαρακτηριστικά ή κάποια σύνδεση να είναι τόσο σημαντικά που παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. Μπορεί επίσης να συναυθεί ότι η σημαντική διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά ενός προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια που παιζουν σημαντικο ρολο στην αποφαση του μπορει επισης να συναφθεί οτι η σημαντικη διαφορετικη συνθεση η χαρακτηριστικα ενος προιοντος θα πρεπει να ειναι τετοια που μπορουν να ε, οδηγήσουν το μέσο καταναλωτή να αγοράσει ένα προϊόν ή να το αγοράσει υπό διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, για ουσιαστικά χαμηλότερη τιμή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σωστή εφαρμογή του προτινόμενου άρθρου 6 της οδηγίας, όμως, ε, θα πρέπει να εξηγηθεί ε, στην εξήγηση, στην αιτιολογική σκέψη, στο αιτιολογικό 43, το οποίο μιλάει για εξαιρέσει ε, που οδηγούν στην μη εφαρμογή του άρθρου 6. Το πρόβλημα είναι ότι το προήμιο της πρότασης ε, μιλάει για επιπλέον κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη και τις διοικητικέ αρχές του για την αξιολόγηση μιας παραπλανητικής συμπεριφοράς ε, στην περίπτωση διπλής ποιότητα. Όπως βλέπετε στην παρουσίασή μου, τα προβληματικά κριτήρια είναι ότι Κατά την αξιολόγηση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα του έμπορου, ε, να προσαρμόσει ε, το ε, προϊόν με το ίδιο εμπορικό σήμα στα γούστα της αγοράς λόγω της εποχιακότητας των πρώτων υλών, της διαθεσιμότητάς τους, των προτιμήσεων του καταναλωτή ή ειδικές στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγιεινή και θρεπτική τροφή ε, και το δικαίωμα των εμπόρων να προσφέρουν ε, προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα σε πακέτα, ε, αλλά να έχουν διαφορετικό βάρο ή όγκο σε διαφορετικέ γεωγραφικέ αγορέ. Το νέο άρθρο 6 θέλει όμως να απαγορεύσει οποιαδήποτε θέση στην αγορά ενός προϊόντος που είναι ίδιο με ένα άλλο προϊόν, εάν τα δύο προϊόντα έχουν τελεί ουσιαστικά διαφορετική σύνθεση. Το πρόβλημα είναι ότι στη διπλή ποιότητα ε, αυτά, αυτοί οι θεμητοί παράγοντε, όπω η διαθεσιμότητα, η εποχιακότητα των πρώτων υλών κτλ. κτλ ε, η του καταναλωτή, ε, η, η πιο υγιεινή τροφή είναι το βασικό ε, θέμα για να αξιολογηθεί η διπλή ε, ποιότητα. Μπορούμε να συνάγουμε ότι ότι αυτοί οι θεμητοί παράγοντες που αναφέρονται στο προήμιο της οδηγίας οδηγούν σε παράκαμψη του προτινόμενου άρθρου 6 σε, στις περισσότερες περιπτώσεις που, όπου δεν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία και οδηγούν σε διπλή ποιότητα προϊόντων. Υπάρχει στην, στην ομολογία ότι υπάρχει το θέμα της ασφάλειας δικαίου που είναι βασική αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας και που απαιτεί να έχουμε ξεκάθαρη ασφα... ε, ρητή νομοθεσία, ε, να την καταλαβαίνουν τα άτομα, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και να δρουν αναλόγως. Θα ήθελα να τελειώσω την παρουσίασή μου με δύο συστάσεις. Μια και ο βασικός στόχος της τροποποίησης της ε, οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στον τομέα των προϊόντων διπλής ποιότητας είναι να έχουμε ασφάλεια δικαίου για τις διοικητικές αρχές οι οποίε αξιολογούν ακριβώς αυτή τη διπλή ποιότητα των προϊόντων, οι αναφερόμενες εξαιρέσεις ε, δεν θα πρέπει να μπουν στο προήμιο της πρότασης. Και η πρόταση θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι σε αυτές τι περιπτώσεις ο καταναλωτής θα πρέπει να καταλαβαίνει πολύ καλά ή να ενημερώνεται πολύ καλά για ό,τι κάνει. Αυτή η να ενημερωνεται πολυ καλα για τι κανει αυτη η τροπολογια του άρθρου 6 δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις ε, πρακτικές διπλής ποιότητας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θα ήταν μια τροπολογία της, ε, του λεγόμενου μαυροπίνακα του παρατήματος 1 της οδηγίας και να βάλουμε και ένα άλλο στοιχείο στο μαυροπίνακα των ε, παραπλαντικών εμπορικών πρακτικών. Ε, όταν αξιολογούμε τις διάφορες πρακτικές που αναφέρει ο μαυροπίνακας, οι διοικητικές αρχές δεν θα πρέπει να κάνουν αυτή τη δοκιμή ε, για αθέμητες πρακτικές. Θα πρέπει να υπάρχει ε, η υψηλότερη δυνατή προστασία του καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε πολύ για μια ε, ακριβέστατη παρουσίαση. Πραγματικά θαυμάσια δουλειά κάνατε και σας ευχαριστούμε πολύ και η μελέτη σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερο όχι μόνο από την παρούσα Επιτροπή Αναφορών, αλλά από ολόκληρο το θεσμικό μας όργανο. Θα είναι στη διάθεση παντό ε, να την ε, έχει στη διάθεσή του και να μπορέσει να την ε, μελετήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μπενασί, Παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ε, ε, κυρία Βίτοβα για την ε, μελέτη και για την καθαρή ανάλυση των, του τρόπου που λειτουργεί η οδηγία. Όπως τονίσατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της το ζήτημα της διετής ποιότητας τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως και έχει αναλάβει ε, κάποιες δράσεις και ιδίως έχει καταθέσει νομοθετικές προτάσεις. Το αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Εγώ θα ήθελα τώρα με τη σειρά μου να τονίσω ότι εμείς θεωρούμε ότι εφαρμόζεται ήδη η οδηγία κατά των παραπλανητικών πρακτικών στην κατανάλωση από προϊόντα τα οποία φέρουν επισημάνσεις και από τους παραγωγούς τέτοιων ε, εμπορευμάτων. Η πρόθεσή μας ήταν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εδώ, διότι από τα πιο δύσκολα ζητήματα σε αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι αθέμητες πρακτικές όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Ε, αυτά τα branded products, products ε, δεν περιλαμβάνουν ισχυρισμού που να λένε, τι επισημάνσει δηλαδή, τι ετικέτε του, ότι είναι τα ίδια παντού. Είναι κάτι, ένα υπόγειο μήνυμα το οποίο προωθεί η στρατηγική, η εμπορευματική στρατηγική, η εμπορική μάλλον στρατηγική των παραγωγών. Εμεί το περιλάβαμε αυτό σε μια τροπολογία που κάναμε για την οδηγία. Θεωρούμε πάντω ότι παραμένει αναγκαίο οι πρακτικές αυτές να λαμβάνονται υπόψη όπως και άλλες παραπλανητικές πρακτικές για τους λόγους που εξηγήσατε εσείς. Δεν αρχίζουμε με την υπόθεση ότι οι έμποροι θέλουν να καταστρατηγήσουν την εφαρμοζόμενη νομοθεσία. Θεωρούν και αυτοί ότι πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια, να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Είναι αναγκαίο όμως και οι ίδιοι να μπορούν να προσαρμόζονται στις συνθήκες των τοπικών αγορών. Και γι' αυτό προτείναμε τροπολογία για την οδηγία αθέμητων πρακτικών και βέβαια στις αιτιολογικές σκέψεις τις οποίες εξηγήσατε και εσείς με λεπτομέρεια. Η νομική μας, ε, η νομοθετική μας πρόταση ε, είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων τώρα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα σήμερα το πρωί ψήφισε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Προστασία των Καταναλωτών, ΙΜΚΟ, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα πορίσματα της μελέτης σας και προτείνει οι πρακτικές αυτές να θεωρηθούν αθέμητες σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα γίνεται η πρόταση τώρα να μπουν στο παράρτημα της οδηγίας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη εξετάσεως όλων των περιβαλλουσών συνθήκων των διαφόρων υποθέσεων, αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη οι αρχές επιβολής του νόμου να αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε βάρος των καταναλωτών. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην, στον ακριβή καθορισμό, βλέπει άρθρο 6 της οδηγίας, ή το να μπει στο παράρτημα. Άρα, μια δοκιμασία λιγότερη, ένα τεστ λιγότερο που καλούνται να κάνουν οι αρχές επιβολής του νόμου. Το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε σήμερα το πρωί από την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών και αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους συνομοθέτες να ολοκληρώσουν το έργο τους και αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι να εξετάσουμε και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που διενεργούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την διτή ποιότητα προϊόντων διατροφής, διότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία ήταν να αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία και να αρχίσουν να εξετάζουν την αγορά με, έχοντας στη διάθεσή τους αντικειμενικές πληροφορίες και σε συνεργασία και με τους ενδιαφερομένους εμπόρους. Διότι όπως είπα και πριν δεν ξεκινούμε από την υπόθεση ότι οι έμποροι προσπαθούν ή έχουν την πρόθεση να καταστρατηγήσουν την ομοθεσία. Οι έμποροι οι εταιρείε, δηλαδή θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν στι αγορέ τα προϊόντα τους και βεβαίως να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές και πελάτε τους. Αργότερα έχουμε και παρουσίαση του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την ε, πορεία της έρευνάς ε, τους. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ διότι είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όλα τα θεσμικά όργανα. Όταν άρχισα να το ε, συζητώ το θέμα αυτό, θεωρητικά μεν το κατανοούσα, αλλά στο προσωπικό επίπεδο ε, δεν το καταλάβαινα πολύ καλά. Ε, μετά όμως πήρα ένα χυμό πορτοκαλιού στην Σουηδία, μου άρεσε πολύ. Μετά πήγα στην Ελλάδα και ήταν κατά κάποιο τρόπο την σιρόπι, ήταν γεμάτο ζάχαρη και πολύ λιγότερο περιεχόμενο σε φρούτο. Τι, αγοράζω πορτοκαλάδα ή αγοράζω σιρόπι. Θα πρέπει να είναι το ίδιο αν είσαι ε, ε, Ευρωπαίος πολίτης και επομένως εξορισμού ταξιδεύεις σε διάφορες χώρες, ε, να μην ε, καταστρέψεις και το πρωινό σου πίνοντας ένα σιρόπι αντί για μια πορτοκαλάδα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Όχι. Καλώς. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά. Α, με συγχωρείτε. Ποιος? Επ' αυτού ο κύριος Πέτερ Γιάρ τουλάχιστον να ευχαριστήσω, διότι το έργο μας εδώ ως νομοθετών οφείλεται και στην αλαζονία των παραγωγών. Εδώ και δύο χρόνια εξελίσσεται η συζήτηση αυτή και εγώ έχω πραγματικά αγανακτήσει από την αντιμετώπιση των ε, παραγωγών. Α, μα όχι, λέει, ασχολούμαστε με τις ε, ε, τοπικέ συνήθειε των ε, καταναλωτών κλπ. Και αν θέλουν οι καταναλωτέ μπορούν να κοιτάξουν αυτά ψηλά γραμματάκια στι ετικέτε. Εγώ είπα τότε ότι εάν το προϊόν Α στην Βορειό Ευρώπη θα έχει διαφορετική, ε, διαφορετική γεύση από ότι έχει το ίδιο προϊόν στη, στην, από ότι στην Νότια Ευρώπη. Ε, δεν τα κάνετε όμως αυτά. Και γι' αυτό ε, προκαλείται η αίσθηση ότι μετρούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο νομοθέτης να λάβει μέτρα και βεβαίως να απευθυνθεί και έκκληση στους παραγωγούς. Εάν αλλάζετε την σύνθεση των προϊόντων, να τα εξηγείτε. Να τα εξηγείτε και να τα γράφετε ε, πάνω στα προϊόντα. Ώστε ο καταναλωτής, εφόσον προμηθευτεί κάποιο προϊόν απανταχού του κόσμου να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι αυτό που αγοράζει είναι αυτό που γράφει πάνω. Ελπίζω οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με πραγματικό ε, τρόπο. Δεν, δεν πρόκειται για κάποια ε, λεπτομέρεια. Είναι ένα μέτρο αποκατάστασης εμπιστοσύνης απέναντι στον καταναλωτή. Άλλωστε αποτελεί και μια ιστορία επιτυχίας τη Επιτροπής Αναφορών, διότι εδώ άρχισε η συζήτηση αυτή και εν πάση περιπτώσει καταφέραμε, θα έλεγα μάλιστα μέχρι και αντίθετα και με την ε, βούληση και προσπάθεια τη βιομηχανία να φτάσουμε να ασχοληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιο ο Πρόεδρος Γιούνκερ. Σα ευχαριστώ Πέτερ. Α, αργότερα ο κύριος Τσάκη. Ο κύριος Χολβένη. Όχι, πολύ ωραία το είπατε το όνομα. Αυτό το «ε» το έχετε κι εσείς οι Σουηδοί. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Καλό είναι που εμείς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Εμείς θέτουμε το θέμα. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μιλούμε για ασφάλεια των τροφίμων. Περίπλοκο θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την θέση αυτή. Ευχαριστώ πολύ πάντως για τη μελέτη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε όμως ακριβή δεδομένα. Και να κάνουμε και τη σχετική επικοινωνιακή προσπάθεια. Το ένα είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Το άλλο είναι η ενιαία αγορά. Ασφάλεια τροφίμων και ενιαία αγορά. Η ερευνήτρια είπε πολλές φορές για την επισήμανση, για τις ετικέτες μπορούμε να μιλούμε για περιφερειακές παραδόσεις κλπ. Αλλά όταν έχει την ίδια ετικέτα, το ίδιο προϊόν στην ενιαία αγορά, αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνονται σεβαστά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι αντικειμενικό το κριτήριο. Βεβαίως και πρόκειται για επιχειρήσεις. Και η αποφασία τους είναι αν θα βάλουν περισσότερη ζάχαρη ή όχι και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη. Ας μην είμαστε αφελείς. τελευταίο. Βεβαίως πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε ε, ώστε να πάψει αυτή η ιστορία με τον μαύρο κατάλογο. Να δούμε πώς μπορούν να ενταθούν οι καλές πρακτικές. Εγώ γνωρίζω και κάποιες πρακτικές οι οποίες ήδη έχουν αλλάξει. Δεν θέλω να κάνω τώρα διαφήμιση σε οποιαδήποτε μάρκα, αλλά ε, για τις σοκολάτες Φεραίρο, που πρόκειται για σοκολάτες, σοκολάτες, αυτά τα στρογγυλά σοκολατάκια, ναι. δεν κάνω διαφήμιση προς Θεού, αλλά άλλαξαν τις ετικέτες και πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό το φάκελο και να κρατήσουμε και τη λίστα καλών πρακτικών και τη μαύρη λίστα. Χρειαζόμαστε καλέ πρακτικέ. Α, ναι, αλλά τώρα όμω προκαταλαμβάνεται τη συζήτηση για την επόμενη αναφορά. Α πάμε λοιπόν κατευθείαν στο αναφερόμενο για, το υπαριθμό, για την υπαριθμό 17, ώστε να μπούμε λίγο περισσότερο στην ε, ε, ουσία ω ε, ζήτημα, αφορμή μάλλον για τη συζήτησή μας. Ο κύριος Λάσλο Σιμάντια 370 του 17 και η κυρία Μάια Μανόλοβα, Βουλγαρική ηθαγενεία, η οποία μάλιστα είναι η, βουλγάρα διαμεσολαβήτρια. Καλώς ήρθατε. Θα δώσω σε κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά 5 λεπτά για να κάνουν την σχετική τοποθέτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω ετοιμάσει κάποια εισήγηση επίσημη, απλώ μια ομιλία όσον αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη, αυτόν τον ε, φορέα ε, που εκ μέρου του μιλούμε. Θέλω να σας πούμε ότι από τότε που αρχίσαμε αυτή τη διαδρομή το Μάρτιο του 2017. Σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μας ε, ακούει η Επιτροπή σας που μας ακούτε σχετικά με τις ανάγκες των ε, πολιτών. Έχουμε επομένως και οπότε έχουμε το νόμο. Έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο, ούτω ώστε να ρυθμιστεί η ποιότητα και το περιεχόμενο διαφορετικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω και να υπάρχει κάποιος ε, έλεγχος. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη υπάρχουν ε, τέτοιες, τέτοιοι μηχανισμοί και υπάρχουν και σχετικές δοκιμές. Ε, βέβαια δεν μπορούν οι ξένοι να καθορίσουν τι, το, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Και γι' αυτό βέβαια από την άλλη μεριά θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία αδειοδότησης και έγκρισης για τα εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης, μόνο η αρμόδια αρχή για την αδειότηση θα πρέπει να επιτρέπει να αλλάζει κάποιο προϊόν επειδή ε, η εταιρεία που το κατασκευάζει θέλει να ανταποκρίνεται στα γούστα των καταναλωτών. Είναι παράδειγμα να υπάρξει πολύ πολύ μικρά στοιχεία η σύνθεση του προϊόντος. Εάν αλλάζει η σύνθεση του προϊόντος, ας αλλάξει και η συσκευασία ή το όνομα του προϊόντος. Δεν θα πρέπει η βιομηχανία να κάνει ό,τι να είναι όσον αφορά ακριβώς τη σύνθεση των προϊόντων. Είναι απαραίτητο να το κάνουν αυτό ε, για να περιορίσουν το κόστος. Ο φορέας μας συνεργάζεται με τις ε, ελληνικές αρχές, γι' αυτό και καταγγέλουμε τα όσα προβληματίζουν τον κόσμο. Θα πρέπει να έχουμε πιο στεγανά συστήματα ελέγχου. Ε, βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο ουγγαρέζικο, το πρόβλημα αφορά όλη την κεντρική και Ευρώπη. Όμω λέμε ότι έχουμε μια αγορά που είναι βασικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί αυτά αντιβαίνουν σε μια ελεύθερη αγορά. Ίσως ευκαιρίε, ε, υγιεινή διατροφή. Χρειάζεται επίση η σωστή διατροφή να περνάει και μέσα από την παιδεία θα πρέπει αυτά να τα αναλάβει κάθε κράτος μέλος. Μιλούμε για ισότητα ευκαιριών, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει αυθαίρετη αλλαγή κάποιου τυποποιημένου προϊόντος. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι θέλουν οι καταναλωτές. Αλλιώς να θεωρείται παραποίηση του προϊόντος, να θεωρείται απάτη αυτό που κάνει η εταιρεία που το κατασκευάζει. Άρα τα κρατημέλη να προσπαθήσουν περισσότερο. όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν ε, πρόσβαση στην ίδια ποιότητα ε, όσον αφορά τα ίδια προϊόντα. Να είναι στεγανή οι κανόνες προστασίας του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. And now the Bulgarian Ombudsman, Mrs. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για Μανόλοβα, η διαμεσολαβήτρια της ε, Βουλγαρίας. Уважаеми Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής των Αναφορών. Σας ευχαριστώ πρώτα πρώτα για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω, να σας πω για αυτή την αναφορά του Οκτωβρίου του 18, όπως μου υποβλήθηκε. Και άλλοι συμπατριώτες μου προσυπέγραψαν αυτή την αναφορά για αυτό το πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς για αυτό τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που αφορεί τα, αφορά τα είδη διατροφής. Πρώτη προϊόντα της ίδιας μάρκας που όμως αλλάζουν σύνθεση και ποιότητα ανάλογα με το κράτος που πήρε σε εμπορία. Επί πολύ καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες είναι αυτή η πρακτική πάρα πολύ κοινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως δημοσιολαβήτρια θεωρώ ότι τέτοια πρακτική θίγει τα δικαιώματα πάρα πολύ σοβαρά όσον αφορά τους πολίτες και η σε βασικές αρχές της Ένωσης Αντιβαίνει επίσης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Είναι μια προσβολή της προσωπικότητας, είναι δυσμενής διάκριση και δεν αφορά δυστυχώς μόνο Βουλγάρους ή μόνο μια μικρή κατηγορία πολιτών. όλους τους πολίτες του αλλά και την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Οπότε, εάν συνεχιστεί μια τέτοια πρακτική, υπάρχει η απειλή του να μονιμοποιηθεί το φαινόμενο της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων και δύο μέτρων και δύο σταθμών. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται περί παραβιάσεως του οργανισμού 1169. Αλλά και παρουσιάζεται η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τα δίμετρα και δύο σταθμά στα είδη διατροφής ήταν ένα βασικό σημείο της Βουλγαρικής Προεδρίας το 18 τότε ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ και είχα καλέσει υπουργού, εκπροσώπου θεσμικών οργάνων από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το φόρουμ η Επιτροπή Γιούροβα μας παρουσίασε τις προτάσεις της για του καταναλωτέ. Εκεί προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα μα είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει ε, πρόκειται των δύο και δύο σταθμών και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία για να επιληθεί το πρόβλημα. Είχαμε επίσης και άλλα θετικά βήματα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Είχαμε μια έκθεση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ιστορικής Χώρας του Κοινοβουλίου που συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις της Επιτροπής σας. Είπαμε ότι θα πρέπει να διατεθούν 2 εκατομμύρια ευρώ για απαραίτητες δοκιμές όσον αφορά το πρόβλημα και ότι θα πρέπει τελικά να υπάρξει ενιαία μεθοδολογία για να επισημανθούν οι διαφορές που δημιουργούν τα δύο μέτρα και δύο Ήδη κάποιος βουλευτής το ανέφερε. Τελικά κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι, ε, κάποιες έχουν σταματήσει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Μετά το φόρουμ της Σόβιας έχουν περάσει 9 μήνες. Εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της ε, νομοθεσίας Πάντως, η δέσμη μέτρων της ε, κυρίας ε, Γιούροβα εξετάστηκε από την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς, έγιναν οι συζητήσεις και από ό,τι έμαθα εγκρίθηκε. με 19 ψήφους υπέρ μια αποχή, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να δοθεί μια λύση μέσω της νομοθεσίας για το πρόβλημα. Ελπίζω ότι κατά αυτή τη θητεία το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βοηθήσει για να υπάρξει απαγόρευση των δύο ε, μέτρων δύο σταθμών. Έτσι τώρα, με αυτή την ομοθετική πρόταση, είπαμε ότι μπορεί να υπάρξουν ελαφρές παραλλαγές ελαφρές παρεκκλήσεις από την ε, τέλεια, την πρώτη ποιότητα, αλλά ότι θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση για τα δύο μέτρα δύο σταθμά, αλλά προσοχή αυτό να μην γίνει παραθυράκι. Πώς, πώς θα οριστεί ακριβώς, το, το, το, πώς θα βρεθεί, αν υπάρχει 5% λιγότερο κακάο σε μια πλάκα σοκολάτα. Ε, αυτό είναι σημαντική ή όχι ως παρέκκληση από την γενική πρότυπη ποιότητα. Ας κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να παρακολουθήσει έτσι και να ελέγξει το Κοινοβούλιο του τι θα γίνει με την υλοποίηση αυτών των νομοθετικών ε, ε, αλλαγών που έχουν γίνει. Με τους αδέλφους μου θα συνεχίσω να ζητώ πλήρη απαγόρευση των διαφοροποίησεων που φέρνουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ίσως πρέπει να συγκροτηθεί κάποιο όργανο πανευρωπαϊκό για να ελέγχει. Και να προβλέπονται και κυρώσεις για τους παραβάτες. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, αρκετούς πόρους ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, 11.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Άρα παρακαλείστε όλοι και όλες να είστε πραγματικά συντομότατοι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Περιμένω μια στιγμή να αλλάξουν οι διαφάνειες. Έχω τώρα και την σχετική συσκευή να σας ενημερώσω σχετικά με αυτά που είπε η ε, διαμεσολαβήτρια της Βουλγαρίας για την εναρμονισμένη μεθοδολογία του Κοινού Κέντρου Ερευνών και επίσης για την επικείμενη εκστρατεία δοκιμασιών για να γίνει καλύτερα κατανοητό το πλαίσιο και το μέγεθος του προβλήματος και η διαφορές που φαίνεται πως υπάρχουν στην ποιότητα των τροφίμων. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι ο ερευνητικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ρόλος μας είναι να δίνουμε επιστημονικές συμβουλές σε αυτούς που ασκούν την νομοθετική πολιτική στην Ένωση. Είμαστε ανεξάρτητοι από εμπορικά συμφέροντα, αλλά και ανεξάρτητοι από εθνικά συμφέροντα. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών δηλαδή. Επανέρχομαι στο θέμα της σημερινής συζήτησης. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέπτυξε πέρσι εναρμονισμένη μεθοδολογία ερευνών, ήδη δημοσιεύτηκε αυτή το 2018, αλλά γιατί. Διότι ανακαλύψαμε ότι δεν είναι εύκολο να συγκρίνονται οι διάφορες δοκιμασίες που γίνονται στις διάφορες χώρες μέλη, τα τεστ δηλαδή. Ο λόγος είναι ότι οι χώρες μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες και οι χώρες μέλη επίσης μας ε, διαβιβάζουν διαφορετικά ε, πορίσματα. Άλλες κάνουν χημικές δοκιμασίες, άλλες κάνουν άλλου είδους και ήταν δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα των τεστ που κάνουν οι χώρες μέλη. Γι' αυτό χρειαστήκαμε ενοποιημένα αποτελέσματα και γι' αυτό φτιάξαμε την αρμονισμένη δοκιμαστική ε, μεθοδολογία. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει στις Εθνικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τους επιτρέψει να κάνουν τα τεστ στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά με σύγκριση των προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλες τις χώρες μέλη. Η μεθοδολογία δοκιμασιών προσφέρει κατευθυντήρες γραμμές σε όλα τα στάδια της, ε, της ε, διαδιαγρασίας των δοκιμών με την επιλογή έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι συγκρίνουμε ε, όμοια πράγματα μέσα από τις ε, δοκιμασίες, όλες τις δοκιμασίες δηλαδή, μέχρι και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Όπως είπα, αυτό είναι έτοιμο από τον Απρίλιο 2018. Τώρα, βρισκόμαστε στο στάδιο που δείχνω στη διαφάνεια, δηλαδή είμαστε στη μέση αυτής της Pan-European Testing Campaign. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, χρειάστηκε να ελέγξουμε αν η μεθοδολογία μας όντως ανταποκρίνεται στον στόχο της. Με άλλα λόγια, αν λειτουργεί, αν αποδίδει και ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα ή τα προβλήματα στην πράξη που θα εμφανιστούν στη διάρκεια των ε, δοκιμασιών. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη σκοπιμότητας για την μεθοδολογία που έγινε από Απρίλιο μέχρι Ιούλιο του 2018. Όπως είδατε ελέγξαμε 64 προϊόντα από 38 παραγωγούς με 410 περίπου ε, δείγματα σε ε, Βέλγιο, κάτω χώρες και Γερμανία για, ως αντιπροσωπευτικές για τις δυτικές χώρες, Αυστρία, Ουγγαρία και Σλοβακία, κεντρικής, κεντρο, κεντρικοευρωπαϊκές χώρες δηλαδή, όλα αυτά είναι κωδικοποιημένα στην ε, βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε κάπως τα αποτελέσματά μας. Έχουμε φτιάξει αυτό το ε, σχέδιο, αυτό το πρότυπο και μιλούμε για ακριβώς ίδια προϊόντα. Δηλαδή, ίδια σύσταση και ίδια ε, ετικέτα. Όταν λέμε απλώς όμοια, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, είτε στην επισήμανση, είτε στην λίστα των συστατικών. Και μικρές διαφορές, για παράδειγμα, η γραμματοσυρά, ε, σημαίνω την ετικέτα. Όταν μιλάμε για διαφορετικά προϊόντα, πάντοτε στην ίδιο πίνακα που βλέπετε, μιλούμε για ποιοτικέ διαφορές, στην ε, αναφορά των συστατικών αλλά και διαφορές στην εμφάνιση. Εν ώψη λοιπόν των αποτελεσμάτων μετά από την πρώτη δοκιμαστική φάση θα δείτε στο πράσινο πεδίο 17% 11 δηλαδή προϊόντα, αυτή είναι η αριθμή για τους οποίους μιλούμε, είναι απολύτως ίδια. Η ίδια συσκευασία και ίδια σύσταση. Μετά έχετε το 90% και 2% που είχαν ταυτόσιμη σύσταση αλλά με ίδια ή διαφορετική εμφάνιση. Τώρα στο δεξιό μέρος βλέπετε το 8% όπου ανακαλύψαμε ότι είναι η ίδια η, ε, η εμφάνιση της συσκευασίας αλλά διαφορετική σύσταση. 16% διαφορετικά στη, στην ε, άνω δεξιά ε, μεριά της διαφάνειας με διαφορετική εμφάνιση και με διαφορετική σύσταση. Να τονίσω εδώ ότι αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι τα τελικά πορίσματα. Είναι τα πορίσματα της ε, ε, μελέτης κοπιμότητας. Έχουμε κάνει και... Μάλλον δεν έχει γίνει εδώ η δοκιμή γεύσης. Δεν μπορεί λοιπόν να μεταφερθούν, να μεταφερθεί το περιεχόμενο της διαφάνειας αυτής ε, αυτού, Πού βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε συμφωνήσει με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την τελική σύσταση του καλαθιού και τον αριθμό των προϊόντων. Ζητήσαμε από τις χώρες μέλη που συμφώνησαν να εμπλακούν στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία. Τα, οι 19 χώρες μέλη που βλέπετε στη διαφάνεια να συλλέξουν σχετικές πληροφορίε και να μας τις διαβιβάσουν μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους. Λάβαμε τις πληροφορίε, αυτές, τις αξιολογούμε τώρα, τη συλλογή αυτή δεδομένων το επόμενο βήμα θα είναι να φτιάξουμε ένα κατάλογο των προϊόντων που θα πάνε για ε, δοκιμή γεύσης, πράγματα τα οποία θα είναι ταυτόσιμα στην ε, πρόστια όψη της συσκευασία, αλλά με διαφορετική σύσταση. Θα κάνουμε λοιπόν το sensory testing, δοκιμή γεύσης και θα έχουμε μετά πλέον έτοιμη την τελική έκθεση. Αν χρειάζεστε άλλες πληροφορίες, ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ας δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για να μπορέσουν να ε, παρέμβουν. Ο κ. Τσάκη πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Δεν χρειάζονται μακρές συζητήσει. Εκ μέρους του ΕΛΚ θεωρούμε ότι έχουμε ένα περίπλοκο θέμα μπροστά μας. Πρόβλημα μάλιστα. Βλέπουμε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Υποστηρίζουμε αυτές τις δραστηριότητε, αλλά είναι και ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε τελειώσει την προσπάθεια. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής, υπάρχουν νέες δραστηριότητες που προωθούνται. Γι' αυτό προτείνουμε να κρατήσετε ανοιχτές αυτές τις αναφορές και να στηρίξετε ε, αυτές τις αναφορές ασκώντας πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσετε τον πολιτικό διάλογο ούτως ώστε να βρεθεί μια πραγματική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν τόσο πολύ λακωνικοί όλοι οι ομιλητές. Θα ήταν τέλειο αυτό η φιλή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βίτοβα για τα όσα μας είπε για την έρευνα αυτή και τα συμπεράσματά της. Είμαστε εδώ με την ε, Βουλγάρα Λαβίτρια και ως Βουλγάρα ε, και μέλος και πολίτρια μιας χώρας που πλήττεται από αυτό το φαινόμενο θα ήθελα επίσης να σας πω ότι οι αναφορές αυτές πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές θεωρώ. Επίσης, ε, μια επιστολή ε, προς τις ε, ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών ε, για να τις ενημερώσουμε. Έχουμε τους κανόνες για, και, και την νομοθεσία για τα τρόφιμα και τους κανόνες αυτούς που επανεξετάζονται και αναθεωρούνται τώρα. το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό. Το ανέφερε και ο κύριος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι είναι σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Επομένως, συνάδελφοι, κάνω έκκληση να κρατήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορές. Ευχαριστώ, ο κύριος, ο κύριος Νέκο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον ε, διαμεσολα... Ε, την διαμεσολαβήτρια. Υποστήριζω και εγώ αυτή την πρωτοβουλία. Ε, μάλιστα μίλησα για αυτό το θέμα στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά αυτό το θέμα και Αναφέρω με ικανοποίηση ότι δεν έχουμε σταθεί απλώς σε δηλώσεις, έχουμε κάνει πράγματα. Έχουμε μια νομική πρόταση για αλλαγές στην οδηγία και τροποποίηση της οδηγίας. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Αυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ. Και χαίρομαι που η κυρία Μανόλοπα με υποστηρίζει. Φυσικά θέλουμε καλύτερες δράσεις γιατί οι πολίτες, ειδικά οι πολίτες που προσχώρησαν ε, με τα τελευταία κύματα της, ε, των διευρύσεων, περιμένουν ακριβώς αυτές τις δράσεις ε, εδώ και καιρό. Υπάρχουν τώρα ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσίες και πρέπει να εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ποιος Ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώ, Πρόεδρε, ότι μετά από αυτή τη συζήτηση η Επιτροπή μας θα είναι ακόμα πιο δημοφιλή στη Βουλγαρία. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ στην επικαιρότητα, απασχολεί πολλούς. Θα ήθελα να σας πω και κάτι διαφορετικό που δεν έχω συχνά την ευκαιρία να το πω. Πριν ε, καν συζητήσουμε τις αναφορές αυτές, ε, ήδη πρέπει να σας πω ότι έχουμε πετύχει κάποια αποτελέσματα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνουν ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα ευρωπαϊκά όργανα όταν είναι σαφές το πρόβλημα, όταν είναι καλά διατυπωμένο το αίτημα και όταν υποστηρίζεται το αίτημα αυτό από διάφορα κράτη-μέλη. Είναι εύκολο και φυσικό να ζητήσουμε την παραμονή της αναφοράς αυτής στην επικαιρότητα, να παραμείνει ανοιχτή, παρότι έχουμε επιτυχίες ήδη. Είμαστε στην αρχή της διαδρομής. Είμαι πεπισμένος ότι οι αρχικές αντιδράσεις ότι είναι τεχνικό και περίπλοκο το θέμα και ότι δεν μπορούμε να βρούμε μεθοδολογία για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, αυτές οι δηλώσεις, αυτά τα προβλήματα δεν ακούγονται πια. Αυτά τα επιχειρήματα έχουν ε, εκλείψει. Θέλω επίσης να ζητήσω ξανά να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να στείλουμε σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε ενωμένοι, τους στηρίζουμε, στηρίζουμε τη δράση τους και τον αγώνα τους και ελπίζω να ακολουθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και αυτές τις πρακτικές ε, και να κάνουμε αυτά που κάνουμε σε αντίστοιχες ε, περιπτώσεις ε, για τέτοιες αναφορές. Ευχαριστώ, κύριος Κούτσεφ. Κόβατσεφ. Ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω την πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Στηρίζω την πρωτοβουλία της κυρίας Μανόλοβα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η αναφορά. Και αφορά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε κοινή μεθοδολογία, κοινού ελέγχου. και αυτές να αναφέρονται σε οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία. Και ελπίζω ότι οι συνομοθέτες θα συνεργαστούν ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, ε, να τελεσφορήσει μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που στέλνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ο κύριος Γοπέ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Τηλεγραφικά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να επιμηκύνω τη συζήτηση. Δεν πρέπει να δοθεί εντύπωση ότι αυτό το πρόβλημα αφορά μόνο τη Βουλγαρία. Όχι, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στη Λιθουανία. Υπάρχουν καταχρήσεις από τους βιομήχανους και τις βιομηχανίες. Πριν από λίγα χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε για αυτό θέα. Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την ακρόαση. Πρέπει να συνεχίσουμε στο τέλος του αγώνα. Η επισήμαση θα πρέπει να είναι κατάλληλη των προϊόντων εννοώ. Όμως, δεν μιλάω για τρόφιμα μόνο και για... Υπάρχουν και τα καλλιντικά, υπάρχουν τα καθαριστικά, ε, υπάρχουν ε, ηλεκτρικές συσκευές που είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Όλα τα προϊόντα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Συνοψίζουμε. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε όλοι με, τον ίδιο, με, την ίδια, με μία φωνή, με τον ίδιο τρόπο, να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών ε, από τα 19 κράτη-μέλη, τα οποία θα δοθούν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος δοκιμών. Ε, I that it's an important... Πιστεύω κι εγώ είναι πολύ, ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή ΙΜΚΟ, που είναι Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ε, να ληφθεί υπόψη ότι ψήφισε με ευρύτατη πλειοψηφία για το πακέτο το καταναλωτικό. Νομίζω ότι θα υπάρξει πρόταση προς τους, καταναλωτε... προς τους συντονιστές, ώστε να προχωρήσουμε από κοινού με την ΙΜΚΟ για αυτό το θέμα, για να συνεργαστούμε, να οργανώσουμε μια ακρόαση, ένα εργαστήρι, μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να χυθεί άπλετο φως για το θέμα αυτό. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, νομίζω. Και βεβαίως να είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς θα συνεχίζεται ο αγώνας, η προσπάθεια. Σας ευχαριστώ όλους ε, όσους ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, γιατί είναι τελείως απαράδεκτη κατάσταση, άδικη κατάσταση αυτή που συμβαίνει στην ε, Βουλγαρία. Βλέπω ότι η Επιτροπή ξαφνικά έγινε βουλγαρική όλος διόλου. Με μια φωνή έτσι λιθουανική που ακούστηκε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Συνεχίζουμε έτσι. Σας ευχαριστώ όλους που ταξιδέψατε και είστε εδώ. Κυρίως την, ε, ευχαριστώ την Ευρωπαία, συγγνώμη, τη Βουργουάρα Διαμεσολαβήτρια, που ήρθε στην ε, πόλη μας για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ όλους και καλό ταξίδι στην ε, χώρα σας, πίσω στη χώρα σας. Πάμε τώρα στην Λιθουανία. Είναι το θέμα περιμόν 18 και αφορά την αναφορά 160 του 18 και εν προκειμένου έχουμε να κάνουμε με είδη και γεωργία. Ο κύριος Σεϊμάντας Πρανάουσκας είναι ο Άναφερ, μας έχει επισκεφθεί και παρακαλώ εσείς οι οποίοι φεύγετε από την αίθουσα να το κάνετε με ησυχία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Now I think is the right moment. Please, the floor is yours, Mr. Έχετε το λόγο, κύριε Πρανάουσκας. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Labą dieną visiems. Pirmininkė, gerbiami. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πέρσι, το Συμβούλιο Γεωργίας και Τροφίμων υπέβαλε αυτήν την αναφορά όσον αφορά τις δυσμενείς διακρίσεις βόρας των Λιθουανών στα πλαίσια της ΚΑΠ. 128.000 είναι επιδοτούμενοι και πάνω από 52.000 Λιθουανοί που υπέγραψαν την αναφορά. Όλοι, όλοι έχουν θυγεί από το φαινόμενο αυτό. Είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε όλα τα σχετικά δικαιώματα. Όμως η γεωργία τη χώρα μας φαίνεται ότι είναι πολίτε β' κατηγορίας. Είμαστε στο 80% των αμέσων πληρωμών και όχι στο 100%. Αυτό έχει αποφασιστεί από είχε αυτό υποστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 14-20 από το που λέτε πλαίσιο. Οπότε η, η Λιθουανή γεωργία ενδιαφέρονται να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος, γιατί είναι βιώσιμη γεωργία, θέλουμε να υπάρχει πράσινη πολιτική και έχουμε τον οργανισμό 13-07 του 17. Συγγνώμη, 13-07 του 13 Τότε είχαμε ε, το σχετική πρημοδότηση και όλα τα οικολογικά μέτρα σχετικά με το κλίμα ισχύουν για όλους, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι η ίση εργασία σημαίνει ίση αμοιβή. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Γιώργο μας, γιατί αυτές οι ενισχύσεις είναι 30% λιγότερες σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Αυτό δεν είναι σωστό. Κλίμα και περιβάλλον, τι είναι πιο φτηνά στην Λιθουανία κατά 30%. Η Επιτροπή είπε να υπάρξει σύγκληση στην περίοδο 14-20 και αυτό αφορά αυτό το 90% τώρα που ε, καταβάλλεται, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα ούτε στη Λιθουανία ούτε σε άλλες βαλτικές χώρες. Και γι' αυτό το Συμβούλιο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2013 απεφάσισε επιλέξει να ανέβει ε, το, ποσό το καταβάλουμε στα 196 ευρώ ένα εκτάριο για όλα τα κρατη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο του κανονισμού που αφορά τις ε, άμεσες πληρωμές για περίοδο 14-20 δεν έλαβε υπόψη την προαναφέρει απόφαση του Συμβουλίου. Οπότε το 2020 θα πάρουν οι Λιθουανοί όχι 196 αυτά ευρώ, αλλά 176, ε, δηλαδή 20 ευρώ λιγότερα. Οπότε αυτό παραβιάζει ό,τι έχει συμφωνηθεί, ό,τι ό,τι προβλέπουν όλες οι συνθήκες. Επίσης η πράξη προσχώρησης λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε 100% για όλες τις πληρωμές εμείς οι Λιθουανοί ε, για το 2013. Παρ' όλα αυτά, όμως όλες αυτές οι άμεσες πληρωμές το 2013 ήταν ε, στα 140 τόσα ευρώ ενώ πήραν 280 ε, οι υπόλοιποι ε, Ευρωπαίοι. Και προσπαθούμε να ε, εξηγήσουμε το πώς υπολογίστηκε αυτή η διαφορετική συμπεριφορά. Δύσκολο. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες χειραγωγήσεις. Έτσι δεν υλοποιούνται οι προτάσεις του Συμβουλίου 196 ευρώ Έτσι δεν βοηθάτε η πολιτική για το κλίμα και για το περιβάλλον στην Λιθουανία. Το είχε πει όσον αφορά την κατάσταση της Ένωσης το 2017 ο πρόεδρος Γιούνκερ. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εργαζομένους β' κατηγορίας. Ούτε γεωργούς β' κατηγορίας. Πάνω από 50.000 Λιθουανία προσυπέραψαν την ε, αναφορά και είπαν το πρέπει να κοιτάξετε να δείτε γιατί υπάρχει αυτού του είδου η στρέβλωση του νομισμού όσον αφορά ε, επίση ε, αυτέ τι άμεσε πληρωμέ που είναι μικρότερε στη χώρα μα. Θα πρέπει η Κομισιόνα μετέλθει ό,τι μέσα να μην αγνοεί το πρόβλημα αυτό που επισημαίνουμε. Η στόχη μα είναι η εξή. Πρώτα-πρώτα αυτό ο οικονομικό φάκελο να μα δώσει ε, αυτά τα 196 ευρώ για εκτάριο ε, και οι σχετικές ε, πληρωμές για κλίμα και περιβάλλον θα πρέπει να είναι όσο είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άμεσες πληρωμές επίσης θα πρέπει να είναι ίδιες με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ε, όρο, μέσο όρο χωρίς ε, να υπάρχει αυτή η διάκριση. Αυτό είναι πλέον αφόρητο. Οι Λιθουανοί, Γεωργοί ε, δεν τον έχονται άλλο και θα μετέλθουμε κάθε μέσο κοινωνική δικτύωση και λοιπά για να διαμαρτυρηθούμε πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε εμείς και σας ευχαριστούμε για τις επιπλέον ε, απαντήσεις που στείλατε σε σχέση με την ε, θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, την οποία και τώρα θα στραφούμε. Έχει το λόγο η κυρία Σαρλότ Σόλτ, ε, Σόντ μάλλον. Καλημέρα σας, λέει η κυρία Σόντου. Ήδη τοποθετηθήκαμε όσον αφορά το περιεχόμενο της αναφοράς. ο αναφέρον και τι απάντησε για αυτά που εμείς έχουμε πει. Να κάνουμε μια διάκριση. Πρώτα πρώτα έχουμε το θέμα του πολιτικού προβληματισμού όσον αφορά την κατανομή της στήριξης από κράτος σε κράτος. Και ένα δεύτερο θέμα είναι η υλοποίηση των όσων συμφωνήθηκαν στο παρελθόν και, και το αν αυτή η υλοποίηση γίνεται ορθά. Πρώτα πρώτα επομένω. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν για το πολιτές πλαίσιο 21 με 27 που βρίσκεται επί της τραπέζης και υποσυζήτηση πρόταση προβλέπει διαφορετικά βήματα για σύγκληση υπέρ των Λιθουανών γεωργών. Επίσης, επιτυχάνεται μια ισορροπία, γιατί χρειάζεται αυτή η σύγκληση, και από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές περικοπές για κανένα κράτος μέλος. Η θέση της Λιθουανίας αφορούσε αυτή την πρόταση. Τα ακούσαμε και από τον αναφέροντα ζητούνται περισσότερες άμεσες πληρωμές. Αυτά όλα ελήφθησαν υπόψη. Και όσον αφορά αυτήν την σύγκριση της άμεσες πληρωμές, αυτά ο νομοθέτης θα τα λάβει υπόψη. Γιατί θα προχωρήσουμε για να δούμε πώς θα προχωρήσει μετά το 2020 το πολιτικό πλαίσιο. Για να δούμε τώρα τη δεύτερη κατηγορία θεμάτων, δηλαδή τα ζητήματα υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί για το τι δίνεται στα κράτη-μέλη. Για δούμε. Τι γίνεται με τις άμεσες πληρωμές στα νέα κράτη-μέλη μετά την προσχώρηση της χώρας για άμεσες πληρωμές. Έγινε αυτό και από την άλλη μεριά είχαμε την εξωτερική σύγκληση των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών, κάτι το οποίο αποφασίστηκε στα πλαίσια του πολιτού πλαισίου για την περίοδο 14 έως 20. να αναδείξουμε κάποια στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε καλύτερα. Σύμφωνα με την παλαιότερη κοινή αγροτική πολιτική, είχαμε στήριξη και άμεσες πληρωμές. Αλλά η διάθεση μέλη δεν γινόταν με συγκεκριμένο ποσό αναεκτάριο ε, Οι πληρωμές γινόντουσαν σύμφωνα με τη συνδεδεμένη στήριξη του παρελθόντος που δινόταν για να αντισταθμίσει τις περικοπές στις τιμές που είχαν αποφασιστεί. Άρα, στήριξη τιμής, της μειωμένης τιμής και αντίστοιχη αντιστάθμιση. Οπότε, με αυτή την ε, στήριξη σε κάθε κράτος μέλος, μπορεί κανείς να το υπολογίσει ένα εκτάριο και βέβαια βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα ανά κράτος μέλος. Διαφορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φυσική συνέπεια αυτού του συστήματος υπολογισμού. Και οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών δεν αφορούν μόνο τη διαφορά μεταξύ νέων και παλαιών ή μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μεταξύ όλων των κρατών σημειώνονται διαφορές σαν αποτέλεσμα της κάπου όπως αυτή χαράχθηκε και όπως εξελίχθηκε διαχρονικά και η στήριξη ανά εκτάριο επομένως δεν οδηγεί με τις διαφορές της σε βάσιμες ε, αξιώσεις ε, καταγγελίες δηλαδή. Τώρα για η εξωτερική σύγκληση του πόσα δίνονται για άμεσες πληρωμές για την περίοδο 14 έως 20 με το πολιτές πλαίσιο. Είναι συνεχής η σύγκληση και συμφωνήθηκαν οι αρχές αυτής. Υλοποιήθηκαν με κάποιο είδους ε, πληρωμές και δεσμεύσεις πόρων. Και έτσι υλοποιήθηκαν οι αρχές της σύγκλησης. Αυτό όλα τα λέει ο κανονισμός 13 του 13 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τι έγινε μετά. Αποφάσισε η Λιθουανία να πάει στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και να αφήσει τις πληρωμές, κάτι που το προβλέπει ως επιλογή ο κανονισμός και κάτι άλλο. Αυξήθηκε η γεωργία όσον αφορά την έκταση που καταλαμβάνει στη χώρα. Καλό αυτό. Ούτε πήγαν τα χρήματα στην έψη της Υπέθρο και έγινε και αύξηση της εκτάσεως. Επομένως, ο υπολογισμός ανεκτάριο των πληρωμών και των ενισχύσεων προκύπτει τώρα μικρότερος για αυτούς τους λόγους. Αυτό έγινε παντού, οπότε κανείς ε, μετακινήθηκε από τις άμεσες πληρωμές στην ανάπτυξη της υπαίθρου ως ενίσχυση. Αυτά προβλέπονται είπαμε από τους χρηματοδοτικούς φακέλους όπως βασικά από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Βάζω τώρα τελεία και ξαναγυρίζω στο πρώτο σημείο ότι δηλαδή συζητείτε το επόμενο πολιτές πλαίσιο και βέβαια και συζητούμε και το πώς θα κατανεμηθούν οι άμεσες πληρωμές στα πλαίσια της ΚΑΠ. Μετά το 2020, για την επόμενη περίοδο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επίκαιρο, γιατί είχε ξεκινήσει να συζητείται το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι υποδιαπραγμάτευση και άρα συνδέονται οι συζητήσεις. Ο κ. Ροπέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Το συζητάμε και εμείς το θέμα αυτό πολύ έντονα στη χώρα μου. Και τα θέματα που ακούστηκαν θα πρέπει να επιληθούν το συντομότερο δυνατόν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν υπογραφές. Γιατί θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς 52.000 ανθρώπους. Δεν υπάρχει διερμηνία προς τα αγγλικά. Και η πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή. Πολύ ωραία. Θα επαναλάβω αυτά που είπα. Τώρα με ακούτε? Ακούτε τη διερμηνία? Να επαναλάβω αυτά που είπα. Ευχαριστώ όλους όσους ε, μάζεψαν υπογραφές γιατί θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους παραβιάζονται. 52.000 ε, γεωργούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι ίσως το ίμιση του γεωργικού πληθυσμού της Λιθουανίας. Αν υπήρχε τέτοια πρωτοβουλία, τότε η Επιτροπή μας αλλά και άλλες επιτροπές και άλλοι φορείς που συζητούν ε, τώρα αυτή την ε, αναφορά ε, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Θα ήθελα να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά γιατί νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό. Το διαπιστώνουμε. Στι συζητήσει που γίνονται για το πουδουπού, για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά όλα αυτά που πετύχαμε δεν αρκούν. Διαπιστώνουμε ότι οι γεωργικοί εκμεταλλευτές των βαλτικών χωρών δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικοί και η γεωργία των βαλτικών χωρών δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική. Ε, οι δικοί μας γεωργικοί εκμεταλλευτές έχουν πολλές δυσκολίες για να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους σε διάφορες αγορές. Όταν ε, οι άμεσες πληρωμές είναι χαμηλότερες, οι τιμές που πετυχαίνουν ε, είναι χαμηλότερες και άρα υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης των γεωργών στις χώρες μας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ζητήσουμε άμεσες πληρωμές αποδεκτές, σε ένα αποδεκτό επίπεδο, σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, τιμές που να είναι αντίστοιχες με τα προϊόντα τους. Το θέμα είναι πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα και υπό ποιες συνθήκες. Ναι, ναι, κλείνω πρόεδρε. Νομίζω ότι οι γεωργοί των βαλτικών χωρών ζητούν πράγματα που είναι απόλυτα λογικά. Δεν ζητούν τίποτα παράλογο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε μία απόφαση που λέει ότι οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο ύψος του μέσου ευρωπαϊκού κοινοτικού όρου του 2013. Αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Όταν οι βουλευτές από τις βαλτικές χώρες πρότειναν την επίλυση αυτού του προβλήματος, μας είπαν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι υποδέστερο από το πρόβλημα του Brexit. Τώρα είναι το Brexit αυτό που μας απασχολεί και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τέτοια προβλήματα. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Είμαι σχεδόν εισηγητής για εκθέσεις που αφορούν αυτά τα θέματα και το θέμα του Brexit. Θέλω να ασχοληθείτε με αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό το πρόβλημα διαιρεί την Ευρώπη. Θα στηρίξω αυτή την ε, ε, αναφορά, λέει ο κύριος Μητροφάνος. Ε, όχι μόνο γιατί είμαστε γείτονε. Ε, οι Λιθουανοί είναι αδερφοί μας και φίλοι μας στην ε, Βαλτική. Αυτός είναι ένας λόγος. Αλλά και γιατί και στη Λετωνία, στη χώρα μου, οι δικοί μας γεωργοί βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση σε σχέση με τη θέση που βρίσκ... στην οποία βρίσκονται η γεωργοί στις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω λοιπόν ότι οι δικές μας χώρες υφίστανται αρνητική ε, διάκριση ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές σε σχέση με τις παλιές ευρωπαϊκές χώρες και τους γεωργούς τους. Θα μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, κοινωνική συνέπεια, αν θέλετε, αυτής της διάκρισης που υφίστανται οι γεωργοί των λεγόμενων νέων χωρών της Ένωσης. Ακούσαμε την παρουσίαση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα και έχουμε την ελπίδα ότι στο εγγύς μέλλον θα επιτευχθούν κάποιοι συμβιβασμοί και θα υπάρξει σύγκληση των άμεσων πληρωμών στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα γίνει κάτι τέτοιο. Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η σύγκληση των άμεσων πληρωμών. Πεθαίνει η υπεθρός μας. Ο κόσμος φεύγει, πάει στις μεγάλες πόλεις, πάει στο εξωτερικό. Λόγω φτώχειας φεύγει. Το χωριό μου βρίσκεται 12 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λιθουανία. Πριν από 20 χρόνια είχαμε 25 σπίτια στο χωριό. Τώρα μόνο 5 σπίτια είναι ανοιχτά. Όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι έφυγαν από το χωριό, πήγαν στις μεγάλες πόλεις. Βεβαίω χάρη στην ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωση με τα προγράμματα συνοχής, φτιάξαμε καλούς δρόμους με άσφαλτο και στη Λιθουανία και στη Λετωνία. Αλλά ακούστε να δείτε, αν δεν αλλάξει τίποτα στην Ήπεθρο, μέσα σε 10-20 χρόνια δεν θα έχουν αρκετό εισόδημα οι κάτοικοι της Υπέθρου για να επιβιώσουν. και δεν θα έχει και νόημα να υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι. Ε, δεν θα υπάρχουν αρκετά λεφτά για να κάνουμε τα βελτιωτικά έργα σε αυτού του δρόμου, γιατί δεν θα υπάρχουν αρκετοί φορολογούμενοι να πληρώνουν φόρου. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να γράψουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε να μας πει πόσο γρήγορα θα γίνει η σύγκληση των άμεσων πληρωμών. Είναι και στο χέρι μας να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν με μια σύνοψη. Όπως είπα, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο βρίσκεται σε φάση συζήτησης. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να παρακαλέσουμε την Επιτροπή Γεωργίας, που είναι η νομοθετική επιτροπή του σώματος, να ε, συντάξει μια ακριβέστατη γνωμοδότηση για το θέμα αυτό και μετά ε, θα μπει και στην CCC, της οποίας είμαι πρόεδρος και θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να το συζητήσουμε. Βλέπω ότι οι συνάδελφοί μου νεύουν καταφατικά. Και ο αναφερόμενος ε, χαίρεται. Όσο λοιπόν χαίρεστε εσείς, άλλο τόσο χαίρομαι και εγώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή επιστροφή στην ε, πατρίδα σας και ας προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά. επανερχόμεθα στην Ιταλία, στην ε, ε, αναφορά υπαριθμών 205. Πρόκειται για τον αναφερόμενο κύριο Γκαρντίνη, ο οποίος θα λάβει το λόγο. Η αναφορά 205. Λέγομαι Λουίτζι Γκαρντίνη. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Επιτροπής αυτής που μας συγκάλεσε εδώ. Θέλω να μιλήσω για την φορμαλδεΐδη ε, η οποία ε, ταξινομήθηκε ως καρκινογόνα ουσία 1β. Ε, είναι επικίνδυνη. Ε, εμείς ε, παράγουμε στην περιοχή μας γύρω στα 19 εκατομμύρια τόνους το χρόνο, Formal στη ζώνη μας ε, μέσω της εταιρείας Πομπονέσκο στη Μάντοβα, 6 ε, χιλιόμετρα από την Μάντοβα, ε, παράγει πάνω από το 12% της φορμαλδεΐδης στην Ευρώπη. Μιλάμε για εργοστάσια επικίνδυνα, γιατί χρησιμοποιούν πάρα πολλά χημικά, τα οποία είναι πολύ τοξικά. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείε που παράγουν φορμαλδεΐδη ε, προσπάθησαν να σεβαστούν την περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει, όμως ε, με βάση τα δεδομένα ε, αυτά που έγιναν δεν είναι αρκετά για να προστατεύσουν την υγεία της, των κατοίκων της περιοχής, η οποία περιοχή αντιμετωπίζει μόλυνση περιβαλλοντική, κυρίως τα παιδιά, τα οποία νομίζω ότι είναι πιο ευαίσθητα από το γενικό πληθυσμό. Έχουν γίνει τρει επιστημονικέ μελέτε, υπάρχει μια τέταρτη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, που έχουν δημοσιευθεί σε πολλά, πολύ έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ε, και έχουν και την έγκριση της έδρας επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου της Βερόνης, της Βερόνας ε, και την υπογραφή του Αλεσάνδρου Μάρκον, ε, καθώς και του επιδημιολογικού παρατηρητηρίου, ε, δείξαν, έδειξαν ότι η φορμαλδεΐδη ακόμα και σε χαμηλή δόση μπορεί να αυξήσει πάρα πολλές ε, παιδικές αρρώστιες, κυρίως αναπνευστικές και να προκαλέσει γενοτοξικές βλάβες, αλλίωση του, των κυτάρων του DNA. Πρόκειται για βλάβες που πρέπει να, αντιστραφούν, όμως είναι η πρώτη φάση διαδικασίας καρκενογέννησης. Ε, μην ξεχνάτε ότι η φορμαλδεΐδη έχει ταξινομηθεί από την ΙΑΡΚ ως ε, καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο. πρόσφατα η ε, ATS ε, από τη Λομβαρδία έχει κοινοποίησει κάποια δεδομένα για την περίοδο 2006-2015 για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας στη Βιαντάνα ε, που συγκρίνονται τα στοιχεία τους με κάποιες ε, περιοχές αναφοράς της επαρχίας Κρεμόνα και Μάντοβα. Από αυτή τη σύγκριση βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναφορά σημαντική στατιστικά στην ε, κοινότητα της Βιαντάνα σε ό,τι αφορά κάποιους δείκτες υγείας. Έχουμε καρδιο... καρδιακές αρρώστιες, αναπνευστικές αρρώστιες σε όλο τον πληθυσμό. Έχουμε αναπνευστικές αρρώστιες σε παιδιά 0-14 ετών. Έχουμε αυθόρμητες αποβολές λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Ε, μιλάμε για αρρώστιες που επιβεβαιώθηκαν από μεγάλους και σημαντικούς ιατρικούς κύκλους. στη Βιαντάνα στο, και στο Πομπονέσκο ε, έχουμε συγκέντρωση της φορμαδεΐδης ε, κατά μέσο όρο πιο ψηλή και από την ε, Νέα Υόρκη. Πρόσφατα έγινε μία μελέτη από τον Μάριο Φραντζίνη που χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση για την πρόληψη των όγκων της Γκουαστάλα και έδειξε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση φολμαδεΐδης σε ε, σώματα υδάτινα, ε, δηλαδή σε επιφανειακά ύδατα, ε, λόγω του ότι σειραίουν εκεί βιομηχανικά λίματα. Έχουμε λοιπόν μόλυνση λόγω φορμαλδεΐδης 200.000 τόνους το χρόνο και αυτό επιδεινώνει την ποιότητα ζωής ε, και τη δημόσια υγεία στην περιοχή. Ζητάμε κάποιες, κάποια μέτρα, κυρίως για τα πιο ευάλωτα άτομα του πληθυσμού, ε, τα παιδιά, αλλά και τους εργαζόμενους, αλλά και όλο τον πληθυσμό. Θέλουμε πάρα αυτά να υπάρξουν τα κοινοτικά όρια στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, ε, κάτω από τα 2 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο με βάση τις βέλτιστες περιβαλλοντικές ε, πρακτικές ε, του 2015 ε, στην νομοθεσία 21 κάθος 19 για τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές ιδίως όταν, χτίζονται, όταν κατασκευάζουμε πλαίσια από ξύλο. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές ε, όταν παρασκευάσουμε αυτά τα, τα πλαίσια από ξύλο και να εφαρμόσουμε τις, ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις εκπομπές της χημικής νομος, βιομηχανίας. Ε, να εφαρμόσουμε επίσης το REACH για την φορμαλδεΐδη και το παράρτημα 16 του κανονισμού 1907 του 2006 και την υποχρέωση να αντικαταστήσουμε σε διάφορους παραγωγικούς κλάδους τις επιβλαβείς ουσίες με μη καρκινογόνες ουσίες. Σας έδωσα πέντε λεπτά, χρησιμοποιήσατε έξι, για να δούμε τώρα τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Έτσι μαντεύοντας λίγο το κόστος σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα έπρεπε να αξιολογηθεί η, η έκθεση των κίνδυνων και θα έπρεπε αυτή η αξιολόγηση πριν το 19 να έχει, ολοκληρωθεί. Και επίσης έχουμε και το παράδειγμα 16 που προβλέπει ότι θα πρέπει να έχει υπολογιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 19. Δηλαδή τώρα, για πέστε μας, τι γίνεται με αυτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστούμε και τον ε, αναφέροντα. Πρέπει να τα πούμε σύντομα, οπότε και εγώ θα σας πω αμέσως για την τελευταία σας ερώτηση. Έχουμε το πρόβλημα 15. Προτείνεται σύμφωνα με το REACH σε σχέση με το σχετικό μητρό να έχει ολοκληρωθεί από την ε, Υπηρεσία Χημικών μέχρι τις 30 πρώτου πληροφορίε υπάρχουν, θα έχουν δημοσιοποιηθεί με τις 30 πρώτου και είπαμε ότι αυτός ο περιορισμός θα είναι το καλύτερο μέτρο προστασίας της υγείας από τους κινδύνους της φορμαλδεΐδης. Προστασία των καταναλωτών. Θεωρούμε ότι η βασική πηγή έκθεσης είναι η χρήση κάποιων υλικών, ρετσινών, ρετίνης που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές και άλλα ελάσματα που χρησιμοποιούνται. Προτείνεται μέσα από την υπηρεσία των χημικών ότι εκεί όπου υπάρχει συγκέντρωση της ουσίας πάνω από κάποια όρια να μην χρησιμοποιούνται τα σχετικά υλικά. Αυτό με έναν τρόπο να ισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε τι γίνεται να υπάρξει περιορισμός και των εισαγωγών αυτών των προϊόντων και ο σχετικός φάκελος στο ΡΑΚ και στο ΣΕΑΚ θα αποσταλούν όλα τα στοιχεία. Αυτές οι αρμόδιες επιτροπές θα αξιολογήσουν το φάκελο και θα γνωμοδοτήσουν. Θα κάνουν επομένως την ε, πρόταση για τους σχετικούς περιορισμούς. Αυτά σε ορίζοντα ενός έτους. Άρα τότε θα λάβουμε αυτέ τι ειδικέ επιτροπές την πρότασή τους για τους περιορισμούς και στη συνέχεια εμεί θα νομοθετήσουμε και θα ε, απευθύνουμε την νομοθεσία αυτή στα κράτη-μέλη. Ο συνάδελφο θα ολοκληρώσει. Καλημέρα σας για να συμπληρώσω αυτά που είπε η συνάδελφος από πλευράς Ρίτσου Να σας πω δύο λόγια όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας και την άμεση ισχύ της. Τις οδηγίες που επικαλέστηκε ο αναφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την κατασκευή κάποιων πάνελ από ξύλο. Έχουμε τώρα κάποιους νέους κανόνες για την φορμαλδαίδη, τους περιοριστικούς κανόνες που ακόμη όμως δεν εφαρμόζονται. Θα γίνουν υποχρεωτικοί από τις 24 ενδεκάτου ενεστόδοσέ τους. Άρα από τότε όλες οι που έχουν τέτοια πάνελ από ξύλο θα πρέπει να δουν κατά πόσο οι άδειε που έχουν ε, εάν συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία. Βέβαια, οι εθνικές αρχές μπορούν και νωρίτερα να αναθεωρήσουν τις σχετικές εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί, τις άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί σε αυτές τις εταιρείες, ανάλογα με αυτά τα συμπράσματα που προαναφέρθηκαν. Αυτά για τα πάνελ. Τώρα, για την ε, παραγωγή καθεαυτής της φορμαλδεΐδης υπάρχει εφαρμοστική πράξη της Ένωσης ορίζονται κάποια όρια εκπομπής της ουσίας αυτής. Για οργανικές χημικές ουσίες, αυτά όλα προβλέπονται από το 17, αλλά από τις 7 12 του 21 θα γίνουν αυτά τα όρια υποχρεωτικά. Και εν προκειμένου οι εθνικές αρχές μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή ε, τους σχετικούς κανόνες και νωρίτερα. Βλέπουμε για 2 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Τέλος. Έχουμε ε, κάποιους άλλους κανόνες για το τι γίνεται όταν φορμαδεΐδη χρησιμοποιείται για επικάλυψη επιφανειών ξύλινων. Και εδώ έχουμε όριο εκπομπής 2 μιλιγράμμα ανά μέτρο. Η οδηγία για αυτές τις εκπομπές προβλέπει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν επί τη βάση αυτών των οριακών τιμών της αδειοδοτήσεις. Και σε περίπτωση σημαντικής μόλυνσης μπορούν οι αρμόδιες αρχές να κάνουν πιο αυστηρές αυτές τις οριακές τιμές, δηλαδή κατώτερος. Τώρα για τις οδηγίες που αφορά τις εκπομπές των ε, βιομηχανιών μπορεί κανείς να προσφύγει, μπορεί κάποια βιομηχανία να προσφύγει όσον αφορά την σωστή όχι εφαρμογή του κριτηρίου της σημαντικής ρήπανση, ε, Η δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και τα κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ διάσω αυτή η κατάσταση. Οι δυο μηχανίε. η πρόεδρο. τωρα θα δωσω το λογο στα μελη τη επιτροπή αναφορων και πρωτα την κυρια ευη ευχαριστω προεδρε ειναι πολυ διάσωφτη η κατασταση οι υπογραφοντες μας παρουσιάζουν ένα πρόβλημα που είναι γενικό από τη χρήση της αλλά και το ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και αφορούν την ε, Βιαντάνο, στην, προβίντσα, στην επαρχία της ε, Μάντοβα, όπου μέσα σε μια περιοχή ακτίνας 6, 6 τετραγωνικών χιλιόμετρων παράγεται το 12% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής. Είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση και με βάση τα επιδημιολογικά, όλες τις επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με βάση τις ε, περιβαλλοντικές μετρήσεις ε, στην ατμόσφαιρα και τον αέρα. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, αναφέροντες που ήρθαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χρησιμοποίησαν το εργαλείο της αναφοράς για να μας πούν ποιο είναι το γενικό αλλά και το τοπικό πρόβλημα. Είμαι ικανοποιημένη και από την απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα γιατί πηγαίνει προς την ευκταία κατεύθυνση, δηλαδή να προστατευτούν οι πολίτες, η υγεία τους και το περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες δράσεις και για τον περιορισμό της χρήσης, ε, για τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν φορμαλδεΐδη, για προϊόντα δηλαδή που όλοι εμείς ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε στην Ένωση, στα επιπλά μας Φερπίν, πολύ απλά, αλλά και ε, σε ό,τι αφορά τα νέα όρια, τα οποία ε, θα αφορούν τους ε, ρηπαντές στην ατμόσφαιρα, π.χ. τη φορμαλδεΐδη για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές. Θα πρέπει λοιπόν οι οριακέ τιμέ να γίνουν σεβαστέ το συντομότερο δυνατό από τι τοπικέ αρχέ τη Ιταλία. Ειδικά λόγω τη πολύ δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στην επαρχία τη Μάντοβα και στην Βιαντάνα κυρίω, στην περιοχή τη Βιαντάνα. Προτείνω λοιπόν οι παρατηρήσεις που μας παρουσίασαν εδώ οι αναφέροντας και οι αναφέροντες και η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κοινοποιηθούν στην επαρχία αυτή, εκεί όπου υπάρχουν χημικές ε, βιομηχανίες που παράγουν δέιδη αλλά και στις εταιρείες αυτές που κατασκευάζουν αυτά τα ξύλινα πλαίσια, ε, αλλά και στην ε, περιφέρεια της Λομβαρδίας, η οποία πρέπει να ακούσει το πρόβλημα και να πάρει αποφάσεις. Να υλοποιήσει μάλλον την απόφαση που ελήφθη πρόσφατα που δεν εφαρμόστηκε σε ό,τι αφορά τις οριακές τιμές των ε, βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Να τους, να τους πούμε λοιπόν και ποια ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε για να προστατεύσουμε και να πλαισιώσουμε την παραγωγική διαδικασία. Γιατί δεν πρέπει να τιμωρήσουμε μία ε, περιοχή η οποία φιλοξενεί πάρα πολλές βιομηχανίες. Ε, βιομηχανίες οι οποίες δεν σέβονται τις οριακές τιμές. Επιπλέον έχουμε και νέα στοιχεία που μας δείχνουν ότι είναι σημαντικό να, κάνουν, γίνουν κάποια πράγματα για να προστατεύσουμε κυρίω ευάλωτου πληθυσμού, τα παιδιά κτλ. Αυτό φαίνεται από τι ε, μελέτε. Όλοι πρέπει να δράσουμε μεγάλη υπευθυνότητα για να εξασφαλίσουμε την υγεία ειδικά των μελλοντικών γενιών. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μητροφάνοφς. Ευχαριστώ. Προτριετίας η ταξινόμηση φορμαλιδίδης άλλαξε από τη λίστα των επικίνδυνων ουσιών, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, δυνατότητα πρόκλησης καρκίνου. Από υποψία δηλαδή πήγε, δεν είναι απλώς πλέον ύποπτη, αλλά είναι μεταξύ ύποπτης και βέβαιας καρκινογόνου ουσίας. Χρησιμοποιείται για την ε, επάλυψη ξύλων πλαισίων. Γιατί, γιατί είναι φτηνή η ουσία αυτή. Η διαδικασία αντικατάστασης της επικίνδυνης αυτής ουσίας έχει παγώσει, διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν δραστηριοποιούνται επαρκώς για να πιέσουν την βιομηχανία να αλλάξει την τεχνολογία αυτή και να αντικαταστήσει την φωμαδείδη με άλλες ουσίες οι οποίες ίσως θα είναι πιο ε, δαπανηρές, πιο ακριβές, αλλά δεν θα είναι τόσο επικίνδυνες για την υγεία. πολίτες που εκτίθενται στην ουσία αυτή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της πρέπει να προστατευτούν. Δεν έχει φτάσει ακόμα στην ε, δυσμενή φήμη του αμοιάντου, αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις και η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της αυτά, καθώς και τις μελλοντικέ συνέπειες στην υγεία και ιδίως των παιδιών που επηρεάζονται από δυσμενείς επιδράσεις στο γενετικό του υλικό. Έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε τις απαιτήσεις και προτάσεις που περιλαμβάνει η αναφορά. Το πρώτο αίτημα της αναφοράς είναι να εφαρμοστούν αυστηρότατες, αυστηρότερες μάλλον τιμές για τις ε, εκπομπές στην ατμόσφαιρα και ιδίως για την κατασκευή ξύλινων πλαισίων όπου χρησιμοποιείται η φορμαλδεΐδη σύμφωνα με την οδηγία του 2015. Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η διαρκής παρακολούθηση δεν είναι κοινώς αποδεκτή πρακτική εγώ θεωρώ όμως ότι αρκεί αυτό για να ισχυροποιηθεί η απέτηση των αναφερομένων. Έχουμε ξεπεράσει το χρονικό όριο, απαντάει η πρόεδρος. Είναι πολύ επιβαρημένη η μερισσία διάταξη. Πραγματικά έχει γίνει πολύ δύσκολη η διεύθυνση της συζητήσεως με τροφάνος. Ναι, ναι, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, λέει η πρόεδρο. Θα αφαιρέσω, θα διαγράψω από τη λίστα των ε, ομιλητών του δύο τελευταίου. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά, όλοι συμφωνούμε επ' αυτού. Θα στείλουμε στην περιφέρεια της Λομπαρδίας ε, επιστολή και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να συντάξει γνωμοδότηση για λογαριασμό μα. και θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι σημειώνεται κάποια κίνηση στον κλάδο αυτό το θέμα είναι ανοιχτό και πρέπει να ε, το θεωρήσουμε ως καλή ευκαιρία για να σημειωθεί μια στενή και θετική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Λοιπόν, πολύ για τα δύο πρόσωπα που διαγράφω από την λίστα. Έχουμε ωστόσο και άλλες αναφορές, άλλες δύο μάλιστα. Η 19 πρώτα στη σελίδα, μάλλον, είναι αδύνατο, είναι αδύνατο να σας δώσω πάλι το λόγο. Αδύνατο. Ο κύριος Ασένσιο Κονσάλες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Χουάν Χωσέ Ασένσιο και είμαι ο δήμαρχος του Βάγεντε Θαμάνθας. Μικρό χωριό. Ε, πυκνότητα για τον πληθυσμό έχουμε τρεις κατοίκους σε ένα τεχνικό χιλιόμετρο. Και τώρα βρίσκομαι στο κέντρο της Ευρώπης ε, έχουμε τελικά πια 25 κατοίκους. Ε, το πρόβλημα ακριβώ είναι η απερίμωση και ε, ερχόμαστε από την αυτόνομη περιφερειακή περιφέρεια τέλο πάντων την πιο μεγάλη της Ισπανίας Καστίγια και Λεών. Είναι πιο μεγάλη την Πορτογαλία, διπλάσιο της Ελβετίας. Τρεις φορές όσο το Βέλγιο και βλέπουμε ότι αυτοί 7 κάτι για τετραγωνικό χιλιόμετρο ε, αντιστοιχούν στην καστή και και αυτό όμως. Αυτό γιατί από τη δεκαετία του 50 ε, είχαμε ε, αστεφιλία Οπότε γι' αυτό και άλλαξε ο τρόπος ζωής. Ε, κτηνοτροφία, γεωργία. είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημά μας. Αλλά οι ηγέτες της χώρας δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό. Αντίθετα, έχουμε λιγότερους δάσκαλους, χειρότερες κρατικές υπηρεσίες και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφη η περιφέρειά μας. Από τη μια μεριά έχουμε τον Ατλαντικό, από την άλλη την Μεσόγειο. Ε, το κλίμα της ΜΕΝ και της άλλης περιοχής ε, συγκλίνουν εκεί. Ε, έχουμε ένα κομμάτι του Natura 2000 ακριβώς γιατί υπάρχει τεράστια βιοπικιλότητα στην φύση μας και επομένως υπάρχει σημαντική κληρονομιά όσον αφορά τη φύση, ε, το, τα, τα, τα τοπία και έχουμε και κάποια προγράμματα, υποδομές τουριστικές ονομάζονται από την διοικητική περιφέρεια. Και επίσης έχουμε ε, Έχουμε γίνει, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για τουριστικά περίπτερα και γι' αυτό θέλουμε να ζητήσουμε να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οικονομήσει τα αιτήματά μας γιατί είχαμε προβλήματα ότι δεν έχει γίνει τίποτε όσον αφορά το δίκτυο Natura 2000. Ε, η νέα, τα νέα έργα υποδομής είναι πάρα πολύ άσχημα για το τοπίο. Δεν έχουν για τα έργα αυτά που έχουν γίνει διαβουλευτεί με τους εκεί κατοίκους. Δεν προστατεύεται το περιβάλλον με αυτά τα έργα. Φύγεται η Το μόνο το οποίο προσέχουν έτσι με αυτά τα έργα είναι τον τουρισμό. Αλλά και αυτός είναι εκτός κάθε ελέγχου, δεν είναι βιώσιμος. Αυτά τα νέα έργα υποδομής είναι πάρα πολύ άσχημα, βλέπετε πόσο χαλάει το τοπίο, ε, δεν προστατεύεται έτσι το τοπίο όπως προβλέπει το Natura 2000 δεν βελτιώνεται η ζωή των ε, ντόπιων, δεν βοηθούν το να επιστρέψει ο κόσμος στην Ήπεθρο. Οπότε ο κόσμος εγκαταλείπει την Ήπεθρο, γιατί δεν υπάρχουν οι βασικές ε, υπηρεσίες όπως ε, παιδεία, συγκοινωνίες, υγεία, πόσιμο νερό, άρα τα έργα αυτά είναι επιβλαβή και δεν είναι καν μια προτεραιότητα. Και ποτέ δεν έγινε διαβούλευση από την ε, περιφερειακή διοίκηση. Α, αυτό ο τουρισμός είναι κατά του Ευρωπαϊκού Δικτύου, είναι κατά παντός νόμου. Αντιβαίνει στην προστασία της ε, ε φύσης. Έχουμε γεμίσει με εργοτάξια τα οποία συνεχίζονται έτσι ανοιχτά ήδη έχουμε 400 έργα ε, επίσης έχουμε και κάποιο είδους ε, ανάπτυξη μεγάλων μονάδων κτηνοτροφίας που θα γεμίσουν τα σούπερ μάρκετ με κρέας χαμηλής ποιότητας θα πρέπει με διάφορο τρόπο να ενημερωθεί ο κόσμος και έτσι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τον τόπο μας και τους συμπατριώτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι μας δίνουν ακόμα λίγα λεπτά οι διερμηνείς. Ελπίζω, ελπίζω. Πέντε λεπτά, ναι. Σας παρακαλώ όμως να είστε συντομότατοι. Να μιλήσετε όσο γίνεται πιο ελάχιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες για την ε, παρουσίαση των ε, στοιχείων. Η Κομισιόν ανέλησε τα στοιχεία αυτής της αναφοράς. Ωστόσο, πρέπει να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου υποδομών ούτε τα έργα τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται, ε, ποια είναι τα κομμάτια του δικτύου Natura 2000 που επηρεάζονται, ε, εάν έχουν γίνει σεβαστές οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αν δηλαδή έχει γίνει στρατηγική αξιολόγηση του σχεδίου αυτού για την τουριστική ανάπτυξη και για κάθε ένα από αυτά τα έργα αν έχει υποβληθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων τις, στους φυσικούς τόπους του δικτύου Natura 2000, που, όπως ε, προβλέπει και η οδηγία για τα ενδιατήματα, τα φυσικά ενδιατήματα. Η Κομισιόν, λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, αρκετά στοιχεία, δεν μπορεί να παρέμβει ούτε να δώσει συνέχεια σε αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Thank you very much. The floor goes to Mrs. Albiol. Κυρία Αλβιόλ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που έφεραν αυτή την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον αγώνα τους για την διατήρηση του τοπίου στην Καστήλη και Λεόν. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις τώρα, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για αυτά τα έργα. Αυτό το έργο ε, περιβάλλεται από φοβερή σιωπή, από αδιαφάνεια. Ε, οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες. Δεν ξέρουμε για ποια περιοχή, για ποια έκταση, ποια έκταση θα επηρεαστεί. Ε, σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτά τα έργα. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν πληροφορίε. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Θα πρέπει οι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και σε αυτέ τι πληροφορίε. Θα θέλαμε λοιπόν να, ζητήσουμε να σταλεί μία επιστολή για αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις πληροφορίες ούτε εμείς ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, συμμετοχή. Η απουσία πληροφοριών οδηγεί σε απουσία συμμετοχής των φορέων που ενδιαφέρονται. Ζητάμε λοιπόν και τις πληροφορίες και οι πολίτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν για να δώσουν την άποψή τους για αυτό το έργο. Και τέλος, το θέμα των κονδυλίων λείπει η πληροφόρηση, λείπει συμμετοχή. Υπάρχει και το θέμα βεβαίως των κονδυλίων. Μιλάμε για υποδομές που σε κομμάτια του δικτύου Natura 2000. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία φύγεται. Θέλω λοιπόν να ζητήσω να αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και θα θέλαμε να μας δοθούν όλες αυτές οι πληροφορίες από τους αναφέροντες, γιατί προς το παρόν δεν τις έχουμε. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε τους αναφέροντες. Πολύ ανησυχητικά όλα αυτά που μας λένε για την τουριστική ανάπτυξη σε Καστιγιλέων. Πρώτα-πρώτα, έλλειψη ενημέρωσης προς τον κόσμο, προς τις δημοτικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε. Δεν τα ξέρει, άρα δεν ενημέρωσε. ότι αυτή. Επίσης, έχουμε όλες αυτές τις ε, παραβιάσει των κανόνων του Natura 2000. Μα ε, αυτό είναι το, το, το, το, το κόσμημα της Καστιγιλίων, αυτή η περιοχή που τώρα θίγεται. Επίσης, όπω σωστά είπε ο αναφέρον, στην Ισπανία και συγκεκριμένα σε Καστήλη Λεόν, το πρόβλημα είναι αυτή, η απερίμωση της υπαίθρου. Το συζητάμε συνέχεια στο Κοινοβούλιο. Έχουμε και έκθεση για αυτό το λόγο. Μα αυτά τα έργα δεν θα κρατήσουν τον κόσμο. Άρα έχουμε όλα αυτά τα τρία προβλήματα. Natura 2000, ε, έλλειψη διαφάνειας, απερίμωση. Ε, για όλους αυτούς τους λόγους στείλαμε επιστολές σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Ούτε καν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενημέρωσαν. Άρα θα πρέπει να δούνε το πώς και θα σβαστούν το 2000 και πώς θα βρουν κάποιο βιώσιμο τρόπο να κρατήσουν τον κόσμο στην Ήπετρο. Η Πρόεδρος. Είναι σαφέστατη η υπόθεση αυτή. Ούτε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκής... Ε, πληροφορίες. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε ανοιχτή την ε, ε, αναφορά, να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τον διάλογο με την χώρα μέλος και τις εθνικές αρχές της και από τη δική μας πλευρά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε επιστολή στην ε, περιφέρεια Καστίδης και Λεών να ρωτήσουμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση και επίσης εάν έχει δοθεί ε, ανώτερη έγκριση ε, γιατί ε, κανείς φαίνεται, δεν φαίνεται να ξέρει ακριβώ. Και μετά θα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ο αναφερόμενος συμφωνεί. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ωραία. Σας εύχομαι λοιπόν καλή όρεξη. Ευχαριστεί η πρόεδρος και τους διερμηνείς που έμειναν ε, λίγα λεπτά παραπάνω και δούλεψαν καλά. Και επανερχόμεθα στις 2.30 στην παρουσία